Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Ελπίζω να φέρατε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας γιατί προβλέπετε αρκετά ε, μεγάλη χρονοβόρα διαδικασία ψηφοφορίας. Κάρμεν την ξέχασες. Everyone Έχετε όλοι μαζί σας τις κάρτες. Δεν έχουν έρθει όλοι όμως αλλά πρέπει να αρχίσουμε. We are on... Πρώτο σημείο της ψηφοφορίας, το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Μπορείτε να περιμένετε δύο λεπτάκια. Έρχεται η Λόρα, αλλά <laughs> κόλλησε στο σανσέρ. Ούτως ή άλλως θα δίνω πρώτα το λόγο στην Ιζαμπέλα, αν θέλει κάτι να συμπληρώσει. Ιζαμπέλα, μπορείς να μιλήσεις μέχρι να έρθουν όλοι οι σοσιαλιστές. Πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω λοιπόν, παίρνω το λόγο. Ε, η αλλως θα δινω πρωτα το λογο στην ιζαμπελα αν θελει κατι να συμπληρωσει ιζαμπελα μπορεις να μιλήσει αφορά τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και ευελπιστώ ότι θα έχουμε πολύ καλή ψηφοφορία. Και εγώ παρατήρησα την κακή λειτουργία των ασανσέρ σήμερα. Γι' αυτό, Πρόεδρε, αν μπορούσαμε να περιμένουμε ένα-δύο λεπτά μέχρι να καταφτάσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, θα ήταν ευχή έργων. <laughs> Συνήθως ε, χαίρομαι όταν ε, είστε λακωνικοί, αλλά αυτή τη φορά δεν μα εξυπηρετεί. Πρέπει να περιμένουμε δύο λεπτά ακόμη. Everybody else is here, so I'm afraid we have to go. Έχουν έρθει όλοι οι υπόλοιποι. Φοβάμαι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Αρχίζουμε. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Α, συγγνώμη, απο, η πρώτη εγκρίθηκε, η δεύτερη απορρίπτεται. Ε, λίγη η ψηφοφορία για την τροπολογία 14. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα ε, με το μηχάνημα. Με τις οθόνες. Λοιπόν, η 13 έχει εγκριθεί. Η 14 είναι που απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται, λέει ο Πρόεδρος. Η ισοπαλία, άρα απορρίπτεται. Σε λάθος οθόνη κοιτάω, λέει ο Πρόεδρος. Amendment rejected. rejected. Απορρίπτεται. Okay, amendment Τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Άρχεται η ψηφοφορία. 37. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται και αυτή. Συμβαστική τροπολογία 4, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 40, γυρίζουμε σελίδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είκοσι ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. πέντε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αιτιολογική ένα 1β νέο, δύο τροπολογία, Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τρία τροπολογία τρία. άρχεται ψηφοφορία. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρχεται η ψηφοφορία για το 5. Ε, ε, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Έχουν ξεπεράσει. Α, εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 23, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9 για την αιτιολογική σκέψη 2. Τροπολογία 9 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Amendment 25. 25 τροπολογία, λέει ο πρόεδρος. Άρχιτη ψηφοφορία. Τροπολογία 25. Τέλο ψηφοφορία εγκρίνεται. Amendment. Τροπολογία 12, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 27, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Amendment 29, the vote open. Ε, απορρίπτεται 29, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται και 32, τελευταία τροπολογία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, σχέδιο νομοθετικής πρόταση. όπως έχει τροποποιηθεί, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται η νομοθετική πρόταση και το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτό. Και συγχαρητήρια στην Ιζαμπέλα Λεβίν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 5, μια στρατηγική για την αλία στην Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Εισηγητής Γκουίντο Μιλάνα. Θέλετε το λόγο κύριε Μιλάνα. Ψηφίζουμε κατευθείαν λοιπόν για το σημείο 5. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 16. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 17. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. It's working, no? Non, ah non, parce que non, recommencer. Amendment 18 19. Η 18 έχει ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 20. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22. Vote closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα Τροπολογία 23. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26 ψηφίζουμε τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται 27 ψηφίζουμε τώρα τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 1 ψηφίζουμε Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 έχει καταπέσει, 30 επίσης. Πάμε στην 31. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32. Δεν δουλεύει πάλι.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 Okay, we'll open the vote on 32. Ψηφίζουμε για 32. It is open. Τέλος ψηφοφορίας. Vote. Τέλος ψηφοφορίας. Ah, it's working now. Α, λειτουργεί τώρα. Τέλος ψηφοφορίας. And it's rejected. Απορρίπτεται. Η 34 έχει αποσυρθεί 33. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35. Ψηφίζουμε. Vote closed. Τέλος ψηφοφορίας. Proved. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. We go down to 39. The vote is open. Πάμε στην 39. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 40. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 41 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρινάται. 42 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 43 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 47. Ψηφίζουμε. Τέλος της Εγκρίνετε Εγκρίνεται. 48. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Α, έχει καταπέσει. Α, με συγχωρείτε, έχει καταπέσει. Οπότε ψηφίζουμε την 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 51. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Τρία ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τέσσερα ψηφίζουμε. Τέλος. Απορρίπτεται. Πέντε ψηφίζουμε. Τέλος, ψηφίζουμε. Τέλος, συγγνώμη, εγκρίνεται. Έξι ψηφίζουμε. Τέλος, εγ... εγκρίνεται πρόεδρος. όχι, απορρίπτεται, διορθώνει. Έπτα ψηφίζουμε. Τέλος, απορρίπτεται. Οκτώ έχει αποσυρθεί, συμβιβαστική 3, ψηφίζουμε. Τέλος, εγκρίνεται. Και περνά... Η 9 έχει καταπέσει λοιπόν, η 10 έχει καταπέσει, πάμε στην 11. Ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 12. Τέλος. Εγκρίνεται. 13. Τέλος, ε, γκρίνεται. 14 ψηφίζουμε. Τέλος, εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το νομοθετικό, την νομοθετική πρόταση όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ψηφίζουμε. Το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τώρα. Ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια τον κύριο Μιλάνο. On to item six, which is the proposal for regulation on genetic resources Το σημείο 6 που είναι η ε, ωφέλεια, η κοινή ωφέλεια, η δεδομή της ωφέλειας ε, από τους γενετικούς πόρους. Δεν θέλει κανείς το λόγο, τον άμεση πληροφορία. Τροπολογία 6. Άρχεται. Τροπολογία 6. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέντε άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Το τροποποιηθέν σχέδιο γνωμοδότησης άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ομόφωνα συγχαίρουμε τον κύριο Χάτσον. ναι, nein. Ναι.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 There Ψηφίσουμε, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους και οδησυγητές. Ε, πολλά χρόνια έγινε θαυμάσια εργασία και στον τελικό τριμερή διάλογο για πολλές ώρες. Ευχαριστώ επίσης την Ιρλανδική Προεδρία. Νομίζω ότι εργάστηκαν ε, τρομερά καλά και για αυτήν και για τις άλλες εκθέσεις για την αλληλεία. Εντυπωσιακή από πολλές απόψεις η Προεδρία τους. Χαίρο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι πολλές από τις προτάσεις που υπευλήθησαν από την πλευρά τους υιοθετήθηκαν με θαυμάσιες τροπολογίες από την Επιτροπή μας και την Ολομέλεια. Ευχαριστώ λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις. Είναι μια καλή βάση για την ε, κοινή οργάνωση της αγοράς και για τις οργανώσεις παραγωγών και συνολικότερα για τον κλάδο. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και τις ε, υδατοκαλλιέργειες, ηχθειοκαλλιέργειες που καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Δεν προτείνω να κάνουμε, να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Δεν χρειάζονται συζητήσεις τώρα. Έχει παρέλθει περίοδος για αυτό το θέμα και το επόμενο κοινή αλληλευτική πολιτική. Αλλά εάν θέλει κανείς ε, να σχολιάσει, παρακαλώ. Η Καρθία Ιέρο. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον να εξηγήσω πώς θα ψηφίσω. Όπως ξέρετε είχαν μείνει μερικά θέματα για να δούμε ποια θα ήταν η θέση ως σοσιαλίστρια και σκιώδης. Κάποιες τεχνικές ε, βελτιώσεις ε, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ότι έχουν συμπεριληφθεί πολλά σημαντικά θέματα και θα επιμείνω σε ένα θέμα γιατί είναι πολύ σημαντικό για την οργάνωση αγοράς. Είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξουν οι νέοι επιχειρηματίες και οι γυναίκες. Όλοι όσοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στη θάλασσα, στις ε, υδατοκαλλιέργειες, γιατί χρειάζονται αποφασιστικά μέσα Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά γιατί σε αυτήν τη συγκυρία κρίση που θίγει τόσο πολύ αυτούς τους δύο τομείς είναι πολύ σημαντικές αυτές οι αναφορές στον κανονισμό. Ευχαριστώ λοιπόν εκπεφρασμένα και να πω στο Συμβούλιο ότι και εγώ έχω συμμετάξει σε πολλές διαπραγματεύσεις όχι στο δημόσιο τομέα αλλά στον ιδιωτικό Πιστεύω λοιπόν πως είναι καλό το κείμενο αυτό και θα το στηρίξω. Ο κύριος Γκάλαχα. Σας συγχαίρω πρόεδρε, δεν ψηφίσαμε ακόμη, αλλά θεωρώ ότι θα υπερψηφιστεί η έκθεση. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία που ανταποκρίθηκε στις ε, μεγάλες προσδοκίες που υπήρχαν εργάστηκαν πολύ σκληρά, ε, επίπονα, συνεργάστηκαν μαζί μας, ανταλλάξαμε απόψεις, ήταν ρεαλιστικοί και την επόμενη φορά που θα είμαι σε ένα κατάστημα και θα δω τις ετικέτες θα σκεφτώ αυτά που συζητήσαμε στους τριμερείς διαλόγους. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την συμβολή τους και ευχαριστώ και την Επιτροπή μας. Και εσείς ε, Πρόεδρε, αντιμετωπίσατε τα θέματα αυτά με πολύ μεγάλη δυσία. Σας ευχαριστώ και είναι καλός ιονός για το μέλλον του κλάδου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Γκάλαχερ. Σας ευχαριστώ για τη σκληρή εργασία σας την ευσυνειδησία σας ε, στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Θέλω να συγχαρώ επίσης και τους καταναλωτές, γιατί θα ψηφίσουμε ένα νέο είδος σήμανσης που θα δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές για το πού έχει αλλιευθεί το κάθε ψάρι. Οι ετικέτες λοιπόν αναφέρουν τον τομέα αλίευσης, το σημείο αλίευσης με κατανοητό τρόπο και τη μέθοδο αλίας, ε, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Αυτό θα αυξήσει την ε, συνειδητοποίηση των καταναλωτών, θα τους δώσει και δυνατότητες επιλογής. Όπως είπε και ο κύριος Γκάλαχερ, και εγώ Όποτε θα δω τη σήμανση των προϊόντων αλίας θα σκεφτώ τι δουλειά κάναμε εμεί εδώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Φερέιρα. Ευχαριστώ. Ένα σχόλιο έχω μόνο που ισχύει και για την ψηφοφορία ως, το ως προς το βασικό κανονισμό της ΚΑΠ. Παρόλο που είναι προκαταρκτική αυτή η ψηφοφορία, σκόπιμο θα ήταν, μια και καλούμαστε να ψηφίσουμε στη φάση αυτή τα έγγραφα, καλό θα ήταν να είχαν μεταφραστεί και σε όλες τις γλώσσες. Είναι κρίμα να ψηφίζουμε μόνο με βάση ένα έγγραφο που υπάρχει στα αγγλικά. νομίζω ότι ακόμη και αν δεν υπήρχαν άλλοι λόγοι, το γεγονό έλλειψη το μεταφράσεων είναι αρκετό λόγο για να μην υπερψηφίσω. Ευχαριστώ για την κατανόησή σα. Βεβαίω είναι κρίμα που υπάρχει μόνο στα αγγλικά το κείμενο αυτό. Προσπαθούμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό στο επόμενο θέμα για το βασικό κανονισμό υπό την Ιρλανδική Προεδρία. Αλλά δεν θα ήταν τον ε, υπό την Ιρλανδική Προεδρία να έχουμε όλες μεταφράσεις. Συνήθως ε, βεβαίω το επιδιώκουμε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την ε, κατανόησή σας. Να περάσουμε στην πληροφορία η οποία και άρχεται. The vote. πέρα 20 υπέρ, 1 κατά, 0 αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερος. Τώρα να περάσουμε στον βασικό κανονισμό. Έκθεση της κυρίας Ρόντουστ. Της οποίας και δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερος την Επιτροπή. Ευχαριστώ την Ιρλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο. Όχι μόνο εδώ, ε, τους παρόντες συναδέλφους. Ευχαριστώ και πάρα πολλούς άλλους συναδέλφους πέραν της Επιτροπής ε, Αλίας. Ιδιαίτερα την ομάδα ε, Αλία για το μέλλον. Όλοι όσοι είμαστε εδώ συνεργαστήκαμε, υπήρξαν χιλιάδες τροπολογίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Μέρες, νύχτες ε, χρειάστηκε να κάτσουμε μαζί και όλοι έτσι μάθαμε κάτι. Παρά τις διαφωνίες μας, ε, παρά την υψηλή συναισθηματική φόρτιση, προέκυψε κάτι το πολύ θετικό Και με χαρά σας ενημερώνω ότι την Παρασκευή ομόφωνα, ομόφωνα επαναλαμβάνω, το Κορεπέρ ενέκρινε το κείμενο αυτό. Όλοι όσοι είχαν αμφιβολίες, ακόμη και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, τώρα συμφωνούν με το κείμενο αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε καλύτερη έκβαση. Ευχαριστώ πολύ τους πάντες και ιδιαίτερα, ακόμη πιο ιδιαίτερα, ευχαριστώ όλους μας τους συνεργάτες. Σε όλα τα επίπεδα. Χωρίς αυτούς ποτέ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιτύχει αυτό που επιτύχαμε. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε βουλευτής είναι τόσο καλός όσο οι συνεργάτες του. Τους ευχαριστώ όλους σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα σημαντικό τμήμα της αλυσίδας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε και ευρύτατη πλειοψηφία στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό και ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ κυρία Ρόντουστ. Αλλά και εσάς πρέπει να σας συγχαρούμε γιατί ήταν μία από τις πιο, από τις πιο δυσχερείς αποστολές κατά τη θητεία μας και με πολύ μεγάλη προσοχή οδηγήσατε το θέμα αυτό σε ευτυχή έκβαση που ελπίζω και στην ψηφοφορία μας σήμερα στην ψηφοφορία, δεν βλέπω άλλα σχόλια, να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία, η οποία και άρχεται. Πέρασε. 20 υπέρ, μία ψήφος κατά, 0 αποχές. Ε, συγχαρητήρια κυρία Ρόντουστ. Οπότε, οπότε, περνάμε στο τέλος των ψηφοφοριών και να περάσουμε στο πιο αγαπημένο μας θέμα. Αλλιεύματα βάθους. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Αρσένη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ακούσουμε σήμερα την παρουσίαση της συμπληρωματικής μελέτης ε, επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. A complementary impact assessment. Η συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων περιλαμβάνει πολύ σημαντικά δεδομένα από τις αναφορές εκφορτώσεων και διάφορες πληροφορίες για τις οικονομικές προσπάθειες που κάνουν τα κράτη-μέλη, γεωγραφικές πληροφορίες, καθώς και πληροφορίες από το σύστημα εντοπισμού των σκαφών. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να ακούμε τον εισηγητή μας. Λιγότερε συνομιλίε, παρακαλώ και λιγότερα πηγαδάκια στου διαδρόμου και όσοι θέλουν να αποχωρήσουν αλλά το κάνω χωρίς φασαρία. Συγγνώμη κύριε Αρσένη. Ε, συνηθίζονται αυτά στο κοινοβούλιο. Αυτή λοιπόν η συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας παρέχει πολύ σημαντικά στοιχεία και δίνει απαντήσεις σε πολύ κέρια ερωτήματα. Ο πρόεδρος, σας παρακαλώ θερμά λίγη ησυχία για να παρακολουθήσουμε τον εισηγητή μας. Όπως είπα και προηγουμένως, λέει ο κ. με βάση το πλαίσιο για τα δεδομένα, και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εκφόρτωση, σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, πληροφορίε από το ημερολόγιο πλοίου και το σύστημα παρακολούθηση των σκαφών, μα δημιουργούν μία πλήρη εικόνα για το 2011 με δεδομένα από όλε τι χώρε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία γνωρίζουμε πια με σαφήνεια ότι αυτό που αναφέρεται στην πρώτη μελέτη επιπτώσεων ε, ευσταθεί ότι μόνο το 1,4% δηλαδή του συναντικών ε, εκφορτώσεων της ΝΕΑΦΚ ε, για τα αλλιευτικά είδη βαθαίων υδάτων καλύπτονται. Επίσης, ε, η μόνη περίπτωση που τα παραγαδιάρικα αποκλείονται από τα στοιχεία αφορούν το γραναδιάρο των βράχων που μπορεί να αλλιευθεί και από μεσοπελαγικές τράτες. Κάτι που δεν αλλάζει ούτως ή άλλως από την πρόταση. Οπότε ό,τι μπορεί να αλλιευθεί από τις βυθότρατες μπορεί να λιευθεί και με άλλα λιευτικά εργαλεία που καλύπτονται από την πρόταση. Και μάλιστα η μετατροπή από τις βυθότρατες στα παραγαδιάρικα είναι δυνατή. Και μάλιστα έχουμε και υπολογισμούς του κόστους αυτής της ε, μετάβασης. Και πολλοί μύθοι και φόβοι και ανησυχίες ε, που διέρευσαν και κυκλοφόρησαν ε, για την ε, νομοθετική αυτή πρόταση διαλύθηκαν με τη χθεσινή δημόσια κρόαση και τη συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν διασκεδαστεί όλες αυτές οι αφιβολίες γιατί τώρα μπορούμε να επισέλθουμε στις λεπτομέρειες για το πού ε, μπορεί να εμφανιστεί ένας αρνητικός αντίκτυπος και να τον αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ ε, σωστή η νομοθεσία και νομίζω ότι και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι πιο στοχευμένα. Και ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να μιλήσω για το μείζον θέμα τη αλίευση καρχαριών από τα παραγαδιάρικα. Με βάση ε, τα ημερολόγια πλοίου και το σύστημα παρακολούθηση καφών καθώ και το πλαίσιο για, τις, ε, για τη συλλογή των πληροφοριών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με τα στοιχεία της αποδεικνύει ότι το 81% του παραλιεύματος καρχαρία βαθέων υδάτων γίνεται από βυθότρατες 13% από παραγαδιάρικα και 6% από τα πλάδια. Οπότε έχουμε πολλά στοιχεία πια για να επεξεργαστούμε και είμαι βέβαιος ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαφωτίσει ακόμη περισσότερο την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ. Να δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Καντέλα για να μας κάνει μια ενημέρωση ω προς τη συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων που ακροθυγώ την είδαμε και χθε, αλλά σήμερα θα έχουμε μια πιο πλήρη παρουσίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή τη σύντομη εισαγωγή που μας έκανε. Πολλά στοιχεία λοιπόν περιλαμβάνει η έκθεση. Δεν θα μακρηγορήσω για να μην σας κουράσω. Θα προσπαθήσω ε, να περάσω τις διάφορες διαφάνειες ε, με ταχύ ρυθμό, εμένοντας όμως τα πιο σημαντικά σημεία. Μία σύντομη υπενθύμηση του ιστορικού υπόβαθρου της πρότασης. Ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα της Επιτροπής, ε, της δικής σας Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τέσσερα βασικά σημεία προσπαθήσαμε να καλύψουμε στη συμπληρωματική αυτή μελέτη επιπτώσεων. Το πρώτο αίτημα είναι η συμπερίληψη των στοιχείων από το πρόγραμμα Deep Fishman θα απαντήσω σε αυτό κατά το τέλο τη παρουσίαση. Επίση, η διευκρίνηση τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Χθε, μάλιστα, σα έδωσα κάποιε πληροφορίε για το θέμα αυτό. Θα προσπαθήσω να τι αναλύσω σήμερα. Ζητήσατε και μία ε, ποσοτικοποιημένη παρουσίαση των δεδομένων αντικτύπου και την ποσοτικοποιημένη επίπτωση των προτινόμενων μέτρων. Και μάλιστα όλες αυτές οι προσπάθειες συλλογής πληροφοριών και από το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών αυτό το σκοπό εξυπηρετούν. Και επίσης μας ρωτήσατε αν μπορούμε να αποτιμήσουμε τον κίνδυνο, τον αντίκτυπο της πρώτης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το τελευταίο σημείο. Και μας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών ε, δεδομένων για επιχειρήσεις αλίας που είναι μικρομεσαίες. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες και καλό θα ήταν στο μέλλον να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τέτοιες πληροφορίες. Θα ήταν χρήσιμο τώρα, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Αν δείτε τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνουν τα κράτη-μέλη για τα ελευτικά σκάφη, σε ό,τι αφορά τον ιολόγιο για παράδειγμα, αλλά και στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Βλέπετε το όνομα του σκάφους, ε, τα διάφορα σήματα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διάφορες άδειες ασφα... Ε, αλευτικές άδειες ασφάλεια και το όνομα του πλειοκτήτη. Αλλά αυτό δεν είναι επιχείρηση. Ο πλειοκτήτης δεν είναι κατά ανάγκη επιχείρηση. Ο μονομένος, ένας μεμονωμένος πλειοκτήτης μπορεί να έχει πλοία σε διαφορετικές εταιρείες ή μια εταιρεία να συγκεντρώνει σκάφη πολλών πλειοκτητών. Οπότε μπορούμε να συγκεντρώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πώς από τις επιχειρήσεις αυτές και σε ποιο βαθμό ασχολούνται με την αλληλή ανοιχτή θάλασσα ή βαθέων υδάτων. Δεν είναι δυνατόν να διασταυρώσουμε αυτά τα δεδομένα, γιατί για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να διασταυρώσουμε τις ελευτικές άδειες για ανοιχτή θάλασσα με το όνομα της επιχείρησης στην οποία ανήκει το σκάφος. Και δυστυχώς τέτοιες πληροφορίες μέχρι σήμερα δεν συγκεντρώνονται από τα κράτη-μέλη. Επιπλέον, στην έκθεση έχετε και κάποιες ε, λεπτομέρειες και μία σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προτείνει ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά ο ορισμός αυτός είναι γενικός δεν μπορεί να μεταφερθεί στο, στην Αλία γιατί στην Αλία έχουμε αλλιευτικά σκάφη και μιλούμε για μεγάλα ή μικρά σκάφη, αλλά δεν μιλούμε για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις και ο χαρακτηρισμός, ο ορισμός μάλλον για τα μικρά σκάφη βρίσκεται στην έκθεση αυτή και στην πρόταση του κανονισμού για το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας. Τώρα, Λαμβάνοντα υπόψη τον ορισμό για τα ελευτικά σκάφη, διαπιστώνουμε ότι 80% του ελευτικού στόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρά. Μικρά ελευτικά σκάφη. 26% της αξίας των εκφορτώσεων και 50% του, του θέσεων εργασίας στην Αλία δημιουργούν αυτά τα μικρά σκάφη. Τώρα, περνάω στην ε, ανάλυση των ε, στατιστικών δεδομένων ε, που συγκεντρώθηκαν και από το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών. Σα είχαμε παρουσιάσει τα δεδομένα αυτά και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε αναλύσει και μην ξεχνάτε ότι αυτά τα στοιχεία τα ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη και όπως είπε και ο κύριος Αρσένης, ζητήσαμε τα στοιχεία για μία τετραετία. Αλλά τελικά συγκεντρώσαμε τις πλήρες πληροφορίες μόνο για το 2011 και με αυτό το χρόνο εργαζόμαστε. Έχουμε 40 εκατομμύρια αρχεία για το 2011. 14 εκατομμύρια αρχεία. Τώρα, ε, τι είναι αυτά τα αρχεία. Έχουμε ένα, μια ελευτική εκστρατεία. Έχουμε το όνομα του σκάφου, τη διάρκεια της εκστρατείας, ε, ε, την αλίευση, στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης σκαφών και έχουμε στοιχεία από 4.456 ελευτικά σκάφη, από τα ημερολόγια πλοίου και τα στοιχεία από το σύστημα παρακολούθησης των σκαφών προέρχονται από 2.835 μόνο σκάφη. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Γιατί μέχρι το 2011 τα, 6, ε, κάτω, τα ε, σκάφη κάτω των 15 δεν ε, ε, ε, περιλαμβάνονται στο σύστημα παρακολούθησης σκαφών. Μπήκαν από το 2012 και μετά. Οπότε μέχρι το 2011 συγκεντρώσαμε στοιχεία μόνο από 2.835 σκάφη. Τώρα, έχουμε τα στοιχεία που μας δείχνουν την ποικιλία των αλληλευτικών ειδών που ελιεύονται σε ανοιχτή θάλασσα. Έχουμε 1.116 διαφορετικά αλληλευτικά είδη. Επίσης, κάθε ελευτικό εργαλείο έχει το δικό του κωδικό. Έχουμε 39 διαφορετικούς κωδικούς για ελευτικά εργαλεία στα δεδομένα που συγκεντρώνουμε. Τα ομοδοποίησαμε όμως σε γενικές κατηγορίες, βυθότρατες, μεσοπελαγικές στράτες, παραγαδιάρικα, κιούρτους και απλάδια για να κάνουμε αυτή την ανάλυση. Θα κοιτάξουμε τις διαφάνειες με τους χάρτες στην πρώτη διαφάνεια βλέπετε το λεγόμενο αποτύπωμα των σκαφών που έχουμε στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών από 2.800 και σκάφη. Βλέπετε λοιπόν τα διάφορα σημεία και στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε και τα ιβερικά χωρικά είδωτα. Πάντως κάθε κουκίδα του χάρτη είναι αυτό που λέμε fishing event, Αλληλευτικό γεγονός, δηλαδή εκεί που γίνονται ε, αλλιεύσεις και αλληλευτικών ειδών βαθαίων υδάτων. Συνολικά η Αλή αυτή καλύπτει όλες τις ατλαντικές ακτές με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, υφαλοκρηπίδα, στην Κελτική θάλασσα. Έχουμε και στα διάφορα νησιά του Νότου αρκετές τέτοιες ε, αλλιεύσεις και μεγάλη συγκέντρωση στο Ρόκολ και στο Χάτονγκ Μπάνκ, Δυτική Σκοτία, ε, ένα τμήμα εμπίπτει στην ΕΑΦ και ένα τμήμα σε άλλη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι δύο κουκίδες εδώ είναι στο, στο μέσο τμήμα του Ατλαντικού. Έχουμε δηλαδή αρκετά ευρεία ζώνη αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Προσπαθούμε τώρα να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς τις διάφορες δραστηριότητες αυτές ανά είδος. Ξεκινούμε με το γρεναδιέρο των βράχων. Η αλία του γρεναδιέρου βράχων γίνονται κυρίως στο χείλος της εφαλοκρηπίδας, Χάτον Μπάνκ και Mid Atlantic Ridge. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ στο χάρτη είναι ότι έχουμε χρωματιστούς κώδικες για, τους για τις βυθότρατες και τα παραγαδιάρικα. Βλέπετε λοιπόν με τα χρώματα αυτά τις διαφορές των δύο αλληλευτικών τρόπων. Έχουμε εδώ νότιο-δυτικά της ε, Ισλανδίας περισσότερες αλλιεύσεις με παραγαδιάρικα. Σε ό,τι αφορά το μαύρο σπαθόψαρο, εδώ έχουμε ένα χάρτη που το περιγράψαμε και στη μελέτη επιπτώσεων. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά των παραγαδιάρικων στο νότο, στα νησιά και στην Πορτοκαλική θάλασσα και σε σχέση με την αλία των βυθότρατων στο, των στο βορρά υπάρχουν θα έλεγα πολιτιστικές διαφορές ό,τι αφορά το πώς γίνεται η αλία μαύρου σπαθόψαρου στο βορρά και στο νότο. Σε ό,τι αφορά την ε, μουρούνα, ε, λίγκα, ενδιαφέρουσες και εδώ οι διαφορές, αλλά υπάρχει τεράστια επικάλυψη μεταξύ της αλίευσης ε, της λίγκας που, έχει, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ειδών βαθέων υδάτων, αλλά αλλιεύεται στην υφαλοκρηπίδα από ό,τι βλέπετε. Πολύ συχνά έχουμε και εμφάνιση ε, της μουρούνας όταν γίνεται αλλία βενθοπελαχικών ειδών, αλλά όχι σε μεγάλο βάθος. Και εδώ έχουμε διαφορετικά αλλιευτικά εργαλεία για την αλλία μουρούνας, ένα ευρύ φάσμα αλλιευτικό εργαλείο, υπερέχουν όμως και πάλι εδώ οι βυθότρατες για την αλλία της μουρούνας. Βλέπετε λοιπόν στο μαύρο χρώμα την αλίευση. Τώρα για το πελαγίσιο λιθρίνη. Αυτό είναι ένα είδος που αλλιεύεται κυρίως σε, από τις νότιες χώρες μέλη, κυρίως από την Ισπανία. Οπότε επανερχόμαστε σε μια κατάσταση αλίας κοντά στην υφαλοκρηπίδα δεν έχουμε πολύ βαθιά είδατε εδώ. Και ακριβώς επειδή το είναι πολύ μικρή κουκίδα, κάναμε ένα zoom και βλέπετε εδώ ότι τα, οι αλληλευτικές προσπάθειες στο χείλος της υφαλοκρηπίδας και γύρω από την Ιβηρική Χερσόνησο και το Βυσκαϊκό Κόλπο είναι πολύ μικρή. Η υφαλοκρηπίδα είναι πολύ περιορισμένη. Το εύρος είναι πολύ μικρό και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πρόκειται για αλληλεία στο χείλος της υφαλοκρηπίδας αλλά και πολύ κοντά στην ακτή. Και εδώ έχουμε μικρότερα αλλιευτικά σκάφη που κάνουν στοχευμένη αλία βαθιάς, βαθαίων υδάτων ανοιχτής θάλασσας. Και εδώ έχουμε χρωματιστούς κώδικες για τα αλλιευτικά εργαλεία και βλέπουμε από το μέγεθος ότι είναι σχετικά μικρό το μέγεθος των πελαγίσεων λιθρινιών και φαίνονται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία για στοχευμένη αλία με δίχτυα. Και εδώ έχουμε κάποιες μπλε κοιλίδες που δείχνουν στοχευμένη αλία ή τουλάχιστον πιθανή στοχευμένη αλία με παραγάδια. Στον άλλο χάρτη βλέπετε κάπως καλύτερα την ε, κατάσταση των ακτών της Ιβερικής Χερσονήσου με τα παραγαδιάρικη αλία στο νότιο τμήμα της Χερσονήσου όπου έχουμε ένα παράδειγμα ελέγχου, υπόδειγμα μάλλον ε, ελέγχου και σωστή διαχείριση. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τις ε, ποσότητες ε, αλλιευμάτων που αλλιεύονται με κάθε είδος εξοπλισμού. Βλέπετε ότι μαζί με τις βυθότρατες και τα σειρώμενα δίχτυα που είναι οι συγκεκριμένες στοχευμένες άδειες, τα ποσά, ε, τα, οι όγκοι είναι περίπου το 54%, ενώ οι άλλοι εξοπλισμοί που δεν επηρεάζονται από αυτή την πρόταση ανέρχονται στο 46% συνολικά. Το 54% για το οποίο κάνουμε λόγο εδώ δεν είναι τα λιεύματα που προέρχονται από στοχευμένα σκάφη, αλλά από όλα τα παραγαδιά, τα, τις βυθότρατες. Εδώ λοιπόν έχουμε το πρόβλημα ότι 54% μπορεί να βρεθεί χωρίς δουλειά, υποτίθεται, αλλά αυτό δεν αληθεύει. Έχουμε ωστόσο κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τα ποσοστά σε όγκο για κάθε είδος του καταλόγου του κανονισμού. Γιατί αν δείτε, τα μεγαλύτερα, είναι, ε, τα μεγαλύτερα αλλιεύματα είναι γκρι μετά ελίγκα και μετά έχουμε τα κοκκινογαριδάκια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαλίες το μουγκρί και τα κόκκινο καριδάκια δεν ε, υπόκεινται στο νέο σύστημα. Αυτά δεν μπαίνουν στα τάκ. Το ίδιο και για το γρεναδιέρο των βράχων και το άλλο, ε, το άλλο ψάρι του, των βράχων, το οποίο δεν είναι κομμάτι των ΤΑΚ, αλλά λέγεται πως ε, δεν εκτιμάται ιδιαίτερα εμπορικά, αλλά έχει δυναμικό. Εδώ έχουμε τις πιθανότητες για τα κράτη-μέλη ανάλογα με τα διάφορα βαθύβια είδη. Βλέπετε λοιπόν για το Γρεναδιέρο των Βράχων έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι στα ισπανικά σκάφη, 44%, να ακολουθούν τα γαλλικά με 26%, ενώ οι υπόλοιποι είναι πολύ πίσω και έχουν πολύ μικρά ε, κομμάτια. Για το μαύρο σπαθόψαρο, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, είναι το πρώτο στην ε, Γαλλία και μετά η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγκα ή Μουρούνα. Και εδώ έχουμε την ε, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία. Η Μουρούνα και πάλι προηγείται η Γαλλία. Για το πελαγίσιο λιθρίνη προηγείται η Ισπανία. Σε αυτά εδώ τα γραφήματα τώρα βλέπετε μια άλλη προοπτική ανάλογα με τις διάφορες τα συμφέροντα μάλλον των διαφόρων σημεών. Γαλλία-Ισπανία κυρίως ενδιαφέρονται για μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών ειδών. Δηλαδή τα συνολικά τους αλλιεύματα ε, ε, είναι, αποτελούνται από διάφορες ποικιλίε, ενώ στην Πορτογαλία βλέπουμε ότι στοχεύουν κυρίως σε ένα-δύο είδη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σαφές, για παράδειγμα ήδη αν δείτε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, που ενδιαφέρονται κυρίως για τη Μουρούνα, τη Γερμανία που αφορά τον ε, Κάβουρα Λάσκας που δεν είναι μέσα στα ΤΑΚ, Δανία, οι χώρες της Βαλτικής, Γαρίδες, ε, το Βυθού και οι κάτω χώρες κυρίως ενδιαφέρονται για τον γουρλωμάτι του Ατλαντικού. Εδώ έχουμε τώρα άλλα γραφήματα για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως. Εδώ έχουμε τα έξι βασικά είδη τα οποία ρυθμίζονται από τα ΤΑΚ και που είναι βασικά εμπορικά. Ποιο είναι το μερίδιο των διαφόρων εξοπλισμών σε αυτά τα αλλιεύματα. Λοιπόν, για τον γερναδιέρο των βράχων βλέπουμε ότι το περιμεγαλύτερο τμήμα γίνεται από τις ε, βυθότρατες για τον ε, Μαύρο σπαθόψαρο έχουμε περισσότερο τις βυθότρατες επίσης, ενώ τα παραγαδιάρικα στα νότια ύδατα κυρίως χρησιμοποιούνται από την Πορτογαλία. Μουρούνα, εδώ είναι ένα αλίευμα το οποίο μπορεί επίσης να, το, να αλιευθεί με τα παραγαδιάρικα, αλλά επικρατούν οι βυθότρατες και αν δείτε την κατανομή αυτών, αυτού του αλιεύματος είναι πολύ σημαντικό παραλίευμα στην αλίευση γάδου και άλλων ειδών, οπότε η επικυριαρχία των, της βυθότρατας ε, οφείλεται στο ότι είναι ε, παραλίευμα ε, άλλων βασικών ειδών. Έπειτα η λίγκα. Επίσης αλλιεύεται είδος μουρούνας, αλλιεύεται επίσης περισσότερο από τις βυθότρατος αλλά και από τα παραγαδιάρικα το πελαγίσιο λιθρίνι κυρίως αλλιεύεται με τα παραγαδιάρικα και η μπεριτσίδα επίσης. Να επαναλάβω κάτι που είπα και χθες γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικό. Πρόκειται για τα αναφερόμενα αλλιεύματα στα ημερολόγια των πλοίων. Καρχαρίες ε, βυθού είναι σε μηδενικά τάκ από το 2009, αλλά ο κανονισμός που ισχύει για το 2009 και το 2010 έδινε τη δυνατότητα εκφόρτωσης μέχρι 10% αυτών των καρχαριών ως παραλίευμα. Για το 2011 και 2012 αυτό το επιτρεπόμενο όριο κυρώθηκε και ο κανονισμός έγινε μηδενικός για τα τάκ καρχαριών βυθού. Από το 2011 λοιπόν δεν ήταν δυνατή η νόμιμη εκφόρτωση καρχαριών βυθού. Και ωστόσο τα στοιχεία του 2011 όπως βλέπετε εδώ τα οποία αναφέρουν οι ίδιοι αναφέρουν παραλιεύματα καρχαριών. Νομίζω πως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως πρόκειται για στοιχεία τα οποία ανήκουν σε μια φάση όπου εκφόρτωση των καρχαριών δεν επιτρέπεται και ωστόσο οι αλληλείς τα αναφέρουν. Είναι καλό το ότι έχουμε αυτές τις αναφορές. Τι συνέβη με τους καρχαρίες που αναφέρθηκαν, δεν μπορούμε παρά να φανταστούμε. Υπάρχει απαγόρευση εκφόρτωσης, οπότε μπορεί κανείς να φανταστεί πως είτε απορρίφθηκαν ξανά στη θάλασσα, αλλά μην με ρωτάτε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Πάντως αναφέρονται, τα στοιχεία αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Και Εφόσον πρόκειται για ένα βαθύβιο είδος, τα μικρά λιεύματα μέσω των παραγαδιάρικων μπορεί να σημαίνουν ότι οι αλληλείς που χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό μπορεί να ελέγξουν καλύτερα τα παραλιεύματα καρχαριών από ότι οι βυθότρατες. Και τώρα περνάμε σε μια ανάλυση που είναι κάπως ε, κουραστική, αλλά απαραίτητη νομίζουμε εμείς. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ είναι να υπολογίσουμε ποιο μερίδιο βαθύβιων ειδών, ποιο είναι μάλλον το μερίδιο των βαθύβιων ε, ειδών στις εκφορτώσεις των ε, σκαφών αυτών. Από τη μια πλευρά έχουμε βάλει τις βυθότρατες και τα πλάδια, γιατί εδώ χρειάζεται ειδική άδεια και έχουμε δύο χρόνια από τότε που άρχισε η ισχύ και από την άλλη έχουμε τα, παρα, τα παραγαδιάρικα, τις ε, ε, μεσοπελαγικές στράτες και τους κιούρτους. Τα στοιχεία αυτά είναι, ε, δείχνουν τον όγκο και την αξία. Τι ποσοστό αξίας, τι, πόσα χρήματα δηλαδή αποφέρουν στους αλληλείς που τα αλλιεύουν. Είναι ο μέσος όρος, εδώ έχουμε όλο τον στόλο, ενώ αργότερα θα δείτε ανά κομμάτι. Εδώ λοιπόν συγκρίνουμε το σύνολο, τα, μάλλον τα βαθύβια είδη σε, σε σχέση με το σύνολο. Αν πάρουμε λοιπόν ολόκληρο το στόλο, βλέπουμε ότι οι βυθότρατες και τα απλάδια έχουν γύρω στο 1,5 και 2% όγκο βαθύβιων ειδών κατά μέσο όρο και η αξία είναι περίπου 4%. Ενώ τα παραγαδιάρικα κτλ. Εδώ ε, τα λιεύματα είναι πολύ χαμηλότερα, γύρω στο 1% και κάτω από το 1%, ενώ η αξία τους είναι γύρω στο το 5 και, ε, μεταξύ μάλλον 5 και 7%. Άρα εν γέννη τα παραγαδιάρικα αλλιεύουν λιγότερα ψάρια αλλά βγάζουν περισσότερα χρήματα σε σχέση με τους άλλους εξοπλισμούς. Τώρα αν δούμε τα διάφορα τμήματα του στόλου έχουμε καταρχήν τα πολύ μικρά σκάφη 10 με 12 μέτρα και βλέπουμε ότι τα παραγαδιάρικα από τη μια πλευρά έχουν μερίδια που οι βυθότρατες, συγγνώμη, από τη μια παιδιά έχουν μερίδια τα οποία είναι πολύ μικρό ποσοστό ε, της, ε, ε, των αλλιευμάτων τους, ενώ τα παραγαδιάρικα εδώ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό, μπορεί να φτάσουν και στο 4%. Έχουν δηλαδή υψηλότερο ποσοστό σε όγκο αλλά χαμηλότερο ποσοστό σε αξία, πράγμα που σημαίνει πως το είδος, τα είδη μάλλον που αλλιεύονται εδώ είναι λιγότερο πολύτιμα. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν πιάνουν καλές τιμές. Το δεύτερο κομμάτι που ακολουθεί, δηλαδή τα σκάφη ανάμεσα στα 12 και τα 18 μέτρα μήκος, εδώ οι τράτες και τα πλάδια στην αξία παραμένουν κάτω από το 3% ε, αλλά ε, ε, αντιθέτως σε σχέση με τον όγκο βγάζουν καλά χρήματα. Ο όγκος είναι κάτω από το 1%. Μπορεί να είναι και μισό της του γενικού αλλιεύματος που είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και είναι ενδεικτικό ότι δεν υπάρχει εδώ στοχευμένη αλλία σε αυτό το τμήμα του στόλου. Για τα παραγαδιάρικα Έχουμε εδώ υψηλότερη οικονομική εξάρτηση, διότι η αξία των αλλιευμάτων βαθύβιων ειδών μπορεί να φτάσει και στο 24%. Πολύ σημαντικό τμήμα λοιπόν τους, ε, της ε, απόδοσης αυτών των σκαφών, των παραγαδιάρικων και των μεσοπελογικών τρατών. Πάμε... τώρα στα 18 με 24 μέτρα. Να από τη μία τα στοιχεία για τις στράτες κάτω από 3% δηλαδή και ένα, καταξία 1% κατόγκου, Πολύ υψηλότερο για τα παραγαδιάρικα στοιχεία 5 με 6%. Σκάφη τώρα. Μεγάλα. Έως 40 μέτρα. Τράτες από τη μια μεριά και απλάδια ανάμεσα στο 5 και 6%, γύρω στο 5% αξία, ενώ τα παραγαδιάρικα είναι γύρω στο 4%. Λίγο κάτω. Και πάλι μεγάλη διαφορά μεταξύ όγκου και αξίας. Και τώρα αν περάσουμε στα πραγματικά μεγάλα σκάφη που μπορούν να ψαρέψουν ε, στην ανοιχτή θάλασσα, φτάνουν μέχρι το Χάτον, τη Μέση, ακόμη και στην περιοχή Νάφο μπορούν να ψαρέψουν. Εδώ βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλή η συμμετοχή των παραγαδιάρικων. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τώρα τα στοιχεία για το 2011. Είναι πολύ χαμηλή η ε, συμμετοχή τους. Το πολύ 1,6%. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγάλη συμμετοχή των παραγαδιάρικων. Αλλά οι τράτες, οι τράτες εδώ η αξία των ε, ε, ειδών ε, μεγάλου βάθους είναι πολύ μεγάλη. Είναι λίγο κάτω από το 9% την καλύτερη χρονιά, το 2009. Αυτό είναι το μέγιστο, το μέγιστο ποσοστό στα συνολικά αλλιεύματα για τα, τις στράτες και τα απλάδια. Αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από 10%. Λοιπόν, να πούμε τώρα και ποια, πόσα είναι τα σκάφη. Θέλαμε να δούμε δηλαδή ποιοι θα φυγούν από τις προτάσεις μας. Τι ποσοστό δηλαδή του στόλου θα αφορά αυτή η πρόταση. Που θα πρέπει δηλαδή να τροποποιήσουν τον τρόπο αλίευσής τους ε, για να συνεχίσουν να αλλιεύουν τέτοια είδη βάθους. Σύμφωνα με το Eurostat έχουμε 37.000 579 σκάφη στον Ατλαντικό. Τα σκάφη για τα οποία έχουμε ημερολόγια πλοίου για το 2011 είναι 4.356. 12% δηλαδή του συνολικού Ατλαντικού στόλου έχει ε, αλλιεύματα τέτοιων ειδών, ο, τέτοιου είδους, οποιοδήποτε και μπορεί να είναι ελάχιστο ή πολύ μεγάλο. Αυτό καλύπτει οποιονδήποτε έχει δηλώσει οποιοδήποτε αλλίωμα τέτοιου τύπου, μεγάλου βάθους δηλαδή. Από αυτό το 12%, από αυτό το 12 πόσα είναι τράτες και ε, απλάδια. Είναι ένα στα 3,5. Μόνο ένα στα 3,5 λοιπόν είναι τράτες και απλάδια. Τα υπόλοιπα είναι παραγαδιάρικα, δεν φύγονται. Από, τα 200 περίπου, ε, από τις 200 περίπου τράτες και απλάδια, πια πιάνουν πάνω από ε, ηχθείες πάνω των 100 κιλών. Αν θέλεις ε, να ε, εκφορτώσεις πάνω από 100 κιλά, τότε χρειάζεσαι άδεια. Από τα 1245 κατεβαίνουμε στα 935 σκάφη και από αυτά 300 ε, πιάνουν λιγότερο από 100 κιλά. Από αυτά τα 935 ε, αλλιεύουν και στοχευμένα και ως παραλιεύματα τέτοιου είδους ε, ψάρια. Πόσοι περνάνε το όριο, το όριο του 10% ε, τέτοια είδη, μεγάλου βάθους, είναι 771. Το 1 πέμπτο δηλαδή του συνολικού στόλου που πιάνει τέτοια είδη και 2% του ατλαντικού στόλου από αυτά τα 771 σκάφη. Τα στοιχεία από τα ημερολόγια λένε ότι ε, το πολύ που αλλιεύουν, από ότι όσο αλλιεύουν, το πολύ τρει μέρες πιάνουν τέτοια είδη. Τα στοιχεία αυτά σημαίνουν ότι η τεράστια αλίευση τέτοιων ειδών είναι παραλιεύματα. Άρα δεν τα αφορά τα περισσότερα σκάφη την τεράστια πλειονότητα των σκαφών αυτών η πρόταση αυτή. Εδώ έχουμε τον αριθμό σκαφών που αφορά η πρόταση. Τι τμήμα της δραστηριότητάς τους αφορά επίσης. Αν δεν θέλεις πλέον άδεια για τέτοια ψάρια. Πόσα σκάφη, συγγνώμη, πόσες δραστηριότητές σου θα πρέπει να μετατρέψει σε κάτι άλλο. Για να κάνουμε αυτή την ανάλυση πρέπει να έχουμε το συνολικό αριθμό αλλιευτικών αποστολών για όλο το έτος. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 14 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα εξετάσαμε. Ο αριθμός ε, ταξιδίων για όλα τα σκάφη δεν θα ήταν δυνατόν να ε, συλλεχθεί και να αναλυθεί. Αλλά για να σας δώσουμε μια ιδέα, μελετήσαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου έχουμε τις προφορίες. πόσα ταξίδια αλληλευτικά έγιναν συνολικά. Βασιστήκαμε στα ισπανικά στατιστικά στοιχεία για τον Ατλαντικό. Εδώ συλλέγουν τέτοιου τύπου στοιχεία. Αν πάρουμε λοιπόν τη συνολική δραστηριότητα των σκαφών αυτών, συμπεριλαμβάνοντα και ταξίδια όπου πιάνουν και βυθού και άλλα, αλλά και ταξίδια όπου δεν πιάνουν τέτοια ψάρια, τη συνολική λοιπόν δραστηριότητα, όχι μόνο όταν υπάρχουν τέτοια αλλιεύματα, η στοχευμένη τέτοιου τύπου δραστηριότητα είναι απλώς 2,8% της συνολικής ετήσιας αλλιευτικής δραστηριότητας. Τι σημαίνει αυτό. Αν τα σκάφη αυτά δεν στοχεύουν πλέον τέτοια αλλιεύματα και μετατραπούν σε παραγαδιάρικα που θα είναι μόνο παραλίευμα, θα αλλάξει μόνο κατά 2,8% η δραστηριότητά τους. Έγινε χθες μεγάλη συζήτηση για το πώς θα γίνει μετατροπή σε παραγαδιάρικα. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές απόψεις, ε, διαφορετικά στοιχεία. Εμείς ως Επιτροπή είχαμε πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, ιδιαίτερα για τα καύσιμά τους, καταδεικνύει, η μελέτη λοιπόν αυτών των στοιχείων καταδεικνύει ότι τα παραγαδιάρικα είναι πιο αποτελεσματικά από πλευράς χρήσης καυσίμων και η μετατροπή ε, μια στρατα 35 35-40 μέτρων σε παρακαδιάρικο είναι 300 με 300 με 320.000 ευρώ. Η συζήτηση βέβαια χθε κατέδειξε ένα σημαντικό στοιχείο. Δεν πρόκειται να ε, ναυπηγηθεί εξ αρχής παραγαδιάρικο Ατλαντικού. Δεν μπορεί με τόσο χαμηλό κόστος. Αλλά είναι εφικτό να τροποποιηθεί μια τράτα σε παραγαδιάρικο με τέτοιο περίπου κόστος. Κάτι άλλο. Η πρόταση δεν λέει στους ε, αλείς να μετατρέψετε τα σκάφη σας σε παραγαδιάρικα. Υπάρχουν και άλλες επιλογές. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τράτες μέσου βάθους, για παράδειγμα για τις συναγρίδες. Ή μπορεί να ε, επιχειρήσουν τα αλλιεύματά τους να είναι κοντά στο όριο με κάποια ε, προσπάθεια να αποφύγουν κάποια αλλιεύματα για να συνεχίσουν να αλλιεύουν περίπου όπως και τώρα. Φτάνουμε στο μεγάλο τμήμα της ανάλυσης για τα γεωγραφικά στοιχεία. Εδώ βλέπετε τη μεθοδολογία μας. Όπως σας είπα, ε, σε κάθε στοιχείο έχουμε όλα τα στοιχεία για κάθε αποστολή. Μπορούμε λοιπόν να πάσα στιγμή, μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε πού είναι κάθε σκάφο από αυτά τα 4.000 περίπου ανά πάσα στιγμή και σε ποιο λιμένα επιστρέφουν, ποιο είναι ο βασικός τους λιμένας. Και μπορούμε να υπολογίσουμε και τα στοιχεία των αλευμάτων των σκαφών αυτών και να υπολογίσουμε και ε, τον αριθμό εργαζομένων που έχουν με βάση τις μελέτες για τα διάφορα τμήματα του ε, στόλου με βάση τα στοιχεία DCF. Προσπαθούμε επίσης να δούμε ποια προστιθέμενη αξία προσφέρουν αυτά τα σκάφη στις περιοχές γύρω από το λιμένα τους. Όχι μόνο από την αλλιευτική δραστηριότητα, αλλά και από άλλες δραστηριότητες. Για να διακριβώσουμε αυτά τα αλλιεύματα ε, των ε, ειδών ε, μεγάλου βάθους, τι προστιθέμενη αξία προσφέρουν σε όλες τις περιοχές προσπαθούμε να καθορίσουμε δύο στοιχεία για κάθε στοιχείο που σας παρουσιάζουμε. Αριθμό σκαφών, εδώ έχουμε δύο διαφάνειες, εδώ βλέπετε το συνολικό αριθμό σκαφών. Παίρνουμε αυτά τα 4.000 σκάφη, 4.400 περίπου, τα παίρνουμε λοιπόν όλα και βλέπουμε σε ποιους ε, λιμένες εκκίνησης ανήκουν. Βλέπουμε που υπάρχουν συγκεντρώσεις, στη Βρετάνη, εδώ, μεγάλη συγκέντρωση. Κατόπιν είναι η χώρα των Βάσκων. Εδώ ένα λιμάνι στη Γαλλικία και δύο λιμάνια στην Ανατολική Σκοτία που βλέπουν στην ε, Βόρεια Θάλασσα. Θα επανέλθω σε αυτά τα σκάφη. Και η μεγαλύτερη συγκέντρωση, η μεγαλύτερη κουκίδα, 44 με 90 σκάφη, εδώ, σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη Βρετάνη, άμα θεωρήσουμε ότι είμαστε στο υψηλότερο σημείο, είναι περίπου 90 λοιπόν σκάφη, εφόσον το πλαίσιο είναι 44 με 90, που είναι και σκάφη που κάνουν στοχευμένοι και σκάφη που κάνουν ε, παρελίευση από αυτά τα είδη. Όλα αυτά τα σκάφη έχουν δηλώσει σε κάποιο σημείο πάνω από 10% αλλιεύματα αυτού του είδου. Εδώ είναι περίπου η ίδια η συμμετοχή αυτών των ειδών, αλλά τα στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά. Η μεγαλύτερη κουκίδα για ορισμένα λιμάνια είναι περίπου 36 με 84 σκάφη. Λιγότερο πλαίσιο δηλαδή. Και εδώ βλέπουμε ότι η συγκέντρωση των στοχευμένων, των σκαφών δηλαδή που κάνουν στοχευμένη αλίευση, είναι μεγαλύτερη στο νότιο τμήμα της Ιρλανδίας. Εδώ ένα μεγάλο τμήμα στοχεύει στην αλίευση τέτοιων ειδών. Κατά τα άλλα, εδώ έχει πολλές μικρές κουκίδες. Πρόκειται για ένα έως τέσσερα σκάφη. Εδώ και σε αυτό το τμήμα της βόρειας Ιρλανδικής θάλασσας, καθώς και στην ακτή της Ανδαλουσίας και τα νησιά. Πόσες θέσεις εργασίας τώρα. Αν εξετάσουμε όλο το στόλο και αυτούς που στοχεύουν και αυτούς που παρελιεύουν, οποιοδήποτε λοιπόν αλίευμα τέτοιου είδους, πόσες θέσεις εργασίας έχουν επιστρέφοντας ε, στον ε, λιμένα εκκίνησης. Τα σκάφη που πηγαίνουν εδώ, που επιστρέφουν λοιπόν εδώ, στη χώρα των Βάσκων, όλα τα σκάφη περιέχουν μεταξύ 421 και 694 εργαζομένων. Είναι για όλα τα σκάφη είπαμε αυτό και για όλα τα ίδια αλλιευμάτων. Δεν είναι οι θέσεις εργασίας που αφορούν μόνο τα ίδια αυτά. Αν δούμε τώρα αυτούς που στοχεύουν σε αυτά τα λεύματα είναι η Σκοτία, η, Σκοτία, η Νοτιωτική Ιρλανδία, η Γαλλικία και λιγότερο στη, Βρετανία στη Βρετάνη και την Ορμανδία. Οι θέσει εργασία αυτές και εδώ αυτές οι θέσει εργασία αφορούν όλα τα λεύματα, όχι τα είδη μεγάλου βάθους. Θα δούμε ε, τις θέσεις εργασίας για τα είδη μεγάλου βάθους, θα τα δούμε αργότερα. Ποσοστό τώρα της απασχόλησης ε, στην περιοχή. Μπορούμε να φτάσουμε στο 19,75% και οι μεγαλύτερες κοιλίδες είναι στη Δανία και τη Γαλλικία. Αλλά αφορούν τα λιμάνια όπου επανέρχονται αυτά τα σκάφη. Συνολικά είναι μόνο μεταξύ 0 και 0,61% της συνολικής απασχόλησης περιοχές αυτές. Η περισσότερη απασχόληση οφείλεται στα είδη μεγάλου βάθους. Όχι. Σε όλα τα λιεύματα που περιέχουν τα σκάφη αυτά. Όχι απλώς τα βυθοπελαγικά. Και αν δούμε τα σκάφη που στοχεύουν σε αυτήν την αλίευση είναι ακόμη μικρότερο το αποτέλεσμα. Αλλά παραμένει υψηλό στη Γαλλικία και τη Δανία στο Κάτεγατ και το Σκάγερακ. Είναι μεγαλύτερες οι κουκίδες εδώ, γιατί είναι μικρότερος ο πληθυσμός στις περιοχές, άρα είναι μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι εξηγείται από το πόσο αραιοκατοικημένες είναι αυτές οι περιοχές. Γι' αυτό είναι υψηλότερο ποσοστό από ό,τι σε άλλες πιο πυκνοκατοικημένες η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Είναι η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχόληση. Εδώ είναι εκατομμύρια ευρώ. Στα λιμάνια όπου η ακαθάριστη η προστιθέμενη αξία είναι μεγαλύτερη, το maximum είναι 6,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η επόμενη τάξη μεγέθους που είναι η πιο συνηθισμένη επίσης είναι ανάμεσα στο 1,5 και 3,8 εκατομμύρια. Εδώ βλέπετε πώς συνδυάζονται σωστά τα στοιχεία. Στους λιμένες της Γαλλικίας είχαμε μεγάλη απασχόληση, αλλά ως ε, προστιθέμενη αξία είναι μικρότερη. Γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον όγκο και την αξία των αλλιευμάτων, ανάλογα με τα τμήματα του στόλου. Πολλά σκάφη στη Γαλλικία, αλλά η αξία των αλλιευμάτων είναι μικρότερη από τα αλλιεύματα στη Σκοτία, την Ιρλανδία, τη Δανία, τη Βρετάνη. Αν εξετάσουμε τώρα τα σκάφη που στοχεύουν αυτά τα διχοπελαγικά είδη στις μεγαλύτερες περιοχές τα μεγαλύτερα ποσά είναι 5,368 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αυτά λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι αναλογίες ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Τι τμήμα δηλαδή της προστιθέμενης αξίας είναι τα βυθοπελαγικά αλλιεύματα. Αν δούμε όλα τα σκάφη, κατά κανόνα, η αξία των βυθοπελαγικών είναι λιγότερο από 1,39%. Αυτή είναι η δεύτερη τάξη μεγέθους που βλέπετε σε αυτές τις κοιλίδες. Αν δείτε τις ε, οθόνες σας, ακόμη και στην Ιρλανδία, τη Βόρεια Σκοτία, τη Γαλλικία, οι κουκίδες αυτές είναι το πολύ 1,39% της ακαθάριστης προσθεθέμενης αξίας για την περιοχή από όλα τα λιεύματα, όλου του στόλου. Η μεγαλύτερη κοιλίδα όπου αυτά τα αλλιεύματα μπορούν να φτάσουν μέχρι 9,27% είναι μόνο στη Δανία. Σε ένα μέρος στη Δανία το ποσοστό είναι ψηλό. Και εδώ είναι περιοχές αεροκατοικημένες και πολύ εξειδικευμένης αλληλείας ίσως. Δεν υπάρχει άλλη οικονομική δραστηριότητα μεγάλης ε, έκτασης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα, τα στοιχεία για, τις, ε, για τη στοχευμένη αλληλεία, βλέπουμε το πολύ 3,71% ε, να είναι το ποσοστό. Πολύ χαμηλό δηλαδή. Και εδώ θα περάσω εντάχει ε, τα τελευταία στοιχεία γιατί τα παρουσιάσαμε εκτενώς την προηγούμενη φορά και ακροθυγώς χθες. Για την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά προορίσματα, σε ό,τι αφορά καταρχήν το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών, ISIS. Βλέπουμε ότι έχουμε δύο αλληλευτικούς πόρους σε καλή κατάσταση, δύο βράχο και μαύρο σπαθόψωρο, σε κακή κατάσταση βαθύβη, βαθύβη οπλώστη, θομπεριτσίδες, μουρούνα και πελαγή λιθρίνι και σταθερή ή χαμηλά φθήνουσα πορεία, το στόκ των σαλούβαρδων και του γουρλωμάτι του Ατλαντικού καθώς και της Λίγκας. Τώρα, άλλα, άλλες συμβουλές της ISIS. βλέπετε εδώ στο link τα πορίσματα που έχουν, που έχουν δημοσιευθεί και η ΝΕΑΦΚ ζήτησε από τη Διεθνέ Συμβούλιο Εξερεύνηση Θαλασσών να, εξερε... να ιδιαίτερα στο θέμα των ε, θαλάσσιων ευάλωτων οικοσυστημάτων και μάλιστα στο Χάτον Bank, στην όχθη Χάτον έχει ε, ερευνηθεί μια περιοχή και θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητη η επέκταση αυτής της ζώνης γιατί παρόλο που είναι μια, ε, μια ζώνη στην οποία γίνεται εκτενής ελεία υπάρχουν μερικά σπάνια είδη ε, και ιδιαίτερα θαλάσσια ε, οικοσυστήματα που εμφανίζονται μόνο σε τρει περιοχέ στον κόσμο. Γι' αυτό προτάθηκε από την ΑΕΣΙΣ κλείσιμο αυτή τη περιοχή ε, του Μπάνκ. Φαίνεται ότι εδώ στην Ευρώπη ε, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο που να χρήζει προστασίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν γνωρίζαμε προηγουμένως που βρίσκονται αυτά τα θαλάσσια, ευάλωτα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Deep Fishman, μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλάβαμε και τα στοιχεία αυτού του προγράμματος και σας τα παρουσιάσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το σχέδιο αυτό συνέβαλε τα μάλα, το Deep Fishman Project, συνέβαλε τα μάλα στη διαχείριση της ανοιχτής θάλασσας, αλλά αφορά κυρίως ε, την επιστήμη των ε, αλληλευτικών αποθεμάτων. Έγιναν εννέα μελέτες ε, για πελαγίσιο, λιθρίνη, μουρούνα, μαύρο σπαθόψαρο και δόθηκα στοιχεία για, το βαθμό αναπαραγωγής αυτών των ειδών, το προσδόκιμο ζωής τους και τις ελευτικές δυνατότητες. Και αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτερα από το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης Θάλασσών και άλλα επιστημονικά σώματα και είναι πραγματικά πολύ καλή συνεισφορά. Γιατί έτσι, ο κλάδος μπορεί με ασφάλεια να, δίνει, να χορηγεί τα στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό και συμβάλλει και στην καλή διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Δεν έχει τόσο σχέση με τα άλλα διαχειριστικά μέτρα και την επιλογή των αλληλευτικών εργαλείων. Σε ό,τι αφορά την Ερμιόνη, το πρόγραμμα Ερμιόνη. Η Ερμιόνη είναι τεράστιο πρόγραμμα. Έγιναν και πολλές δημοσιεύσεις ε, σχετικά και το έργο του προγράμματο Ερμιώνη είναι κυρίως συμβουλευτικό προς το Διεθνέ Συμβούλιο Εξερεύνησης ε, Θαλασσών. Και δίνει στοιχεία για τις βιολογικές κοινότητε ε, στο βαθύ βιοπεριβάλλον, τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά τα βαθύβια οικοσυστήματα, γιατί δεν είναι απλώς ε, αληφτικά πεδία αυτές οι ζώνες, αλλά έχουν και άλλη χρήση. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην καταμέτρηση του ανθρώπινου αντικτύπου και μάλιστα η μελέτη που αναφέρεται εδώ και στην έκθεση δείχνει ότι ακόμη και με τις πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, αν συγκρίνουμε τα σιδερένια, ε, τα τσαλένια καλώδια και ε, τις ε, ε, τους υπολογισμούς ε, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση άνθρακα, τις επιστημονικές έρευνες και τη χρήση των καυσίμων και αν προσπαθήσουμε σε συγκεκριμένες ζώνες να αποτιμήσουμε τον, την επίπτωση αυτών των δραστηριοτήτων, βλέπουμε ότι οι αλληλευτικές δραστηριότητες έχουν, έχουν αντίκτυπο πολύ μεγαλύτερο από ότι ε, όλες οι προηγούμενες δραστηριότητε δραστηριότητες μαζί. Ένα πολύ ενδιαφέρον τμήμα της Ερμιώνης δείχνει ε, κάποια στοιχεία από τη Μεσόγειο. Παρόλο που η Μεσόγειος δεν εμπίπτει στην πρόταση, το έργο της Ερμιώνης, πρόγραμμα της Ερμιώνη για τη Μεσόγειο είναι αξιοσημείωτο, γιατί δείχνει την αληφτική δραστηριότητα σχετικά ρηχά ε, ύδατα σε περιοχές που δεν υπάρχουν κοράλια, αλλά οι τράτες που αλλιεύουν στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι ε, αναδεύουν το βυθό και δημιουργούν ε, ε, ζημιές στα κοράλια που βρίσκονται από κάτω. Δεν είναι ότι ψαρεύουν επί τούτου κοράλια, αλλά είναι ότι καταστρέφουν το, το βυθό. Οπότε και αυτές οι επιπτώσεις θα πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη και για πρώτη φορά το πρόγραμμα Ερμιώνη τη συμπεριλαμβάνει. Το Coral Fish, άλλο σημαντικό σχέδιο και Εδώ επικεντρωνόμαστε σε δύο βασικές μελέτες ε, του Coral του προγράμματος Coral Fish. Το έργο του Coral Fish έγκυται στη συγκέντρωση των στοιχείων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα μας δείχνει ε, σε ποιες ζώνες μπορούμε να βρούμε τέτοια σύβηση, δηλαδή ε, κοράλια ψυχρού ύδατος. Εδώ φαίνεται ότι Έχουμε αρκετές ζώνες με τέτοια κοράλια ψυχροϊδατός και έχουν γίνει και συγκεκριμένες μελέτες για το, την εφαρμογή του κανόνα move on, που δεν είναι και πολύ θετική. Ίσως ε, η Ερμιόνη, ίσως έκανα λάθος εδώ, η Ερμιόνη έδειξε τη σημασία των ε, κοραλιών ε, ψυχρών υδάτων σε ό,τι αφορά το θέμα του, της θέσμευσης άνθρακα. Τώρα, διαδικασία διαβούλευσης. Στο τελευταίο σημείο να σας υπενθυμίσω τα βασικά στοιχεία. Διήρκεσε 18 μήνες ε, από την έναρξη των διαβουλεύσεων μέχρι την κατάθεση της πρότασης, δηλαδή ήταν αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Έγινε διαβούλευση με 12 χώρες μέλη, ε, αυτέ που μα έχουν υποβάλει τα στοιχεία και 5 περιφερειακά συμβουλευτικά, 5 συμβουλευτικές Ζητήσαμε μάλιστα σχόλια από έξι μέλη και δύο ΡΑΚ και μάλιστα είχαμε πολύ τακτικές ε, συνεδριάσεις. Φυσικά οι πόρτες μας είναι ανοιχτές, ε, είναι ευπρόσδεκτοι και εκπρόσωποι του κλάδου και με κυβερνητικών οργανώσεων και μάλιστα είχαμε ειδικέ ε, συνεδριάσεις με τα κράτη-μέλη με θέμα ακριβώς αυτή την πρόταση. Και οι πέντε τελε... επιλογές ε, της πρότασης είναι το καρπός αυτής της διαδικασίας. Ελπίζω με την μελέτη αυτή να δικαιολογούμε, να αιτιολογούμε επαρκώς τα προτινόμενα μέτρα και από το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτά τα μέτρα είναι τα μέτρα που την χάνουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Δεν είμαι υπέρ τη ολοσχερού απαγόρευση, αλλά μια σταδιακή εξάλληψη των επιζήμιων αλληλευτικών εργαλείων. Ο διάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται και είναι σημαντικό και για την Επιτροπή να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και είναι κάτι που μας ενδιαφέρει προκειμένου να έχουμε μια εμπεριστατωμένη απόφαση. Και με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάσαμε και τη συμπληρωματική αυτή μελέτη. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας. Αλλά πραγματικά η έκθεση βρήθη πληροφοριών και τώρα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. ήταν πραγματικά πολύ εκτενή και εμπεριστατωμένη η έκθεση, κυρία Καντέλα. Πέντε ζήτησαν το λόγο ε, ευρωβουλευτέ. Πρώτη, κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Καντέλα. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπε χθε η κυρία Πατράο. Ε, πολύ συχνά αναφέρεται ως παράδειγμα και στην προφορική παρουσίαση και στην έκθεση ε, την Ισπανία ως παράδειγμα, αλλά δεν συμπίπτουν τα στοιχεία που μας δίνετε εσείς από τις Ισπανικές αρχές με αυτά που έχουμε εμείς. Φαίνεται ότι υπάρχουν κενά στην ροή αυτή των πληροφοριών. Και ξεκινώ από τα βασικά στοιχεία της μελέτης, που είναι τα δεδομένα. Είπατε ότι χρησιμοποίησατε δύο είδη δεδομένων από το, γεωγραφικό σύστημα, από το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, από τα ημερολόγια πλοίου και το σύστημα παρακολούθησης ε, σκαφών αλλά αναγνωρίσατε ότι δεν λάβατε υπόψη τα στοιχεία ημερολογίων πλοίου, πλοίων που είναι κάτω των 12 μέτρων, γιατί δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, ούτε λαμβάνετε υπόψη τα σκάφη κάτω των 15 μέτρων, γιατί μέχρι το 2012 δεν ήταν υποχρεωμένο να εμπίπτουν στο σύστημα παρακολούθησης σκαφών. Και μας το αναφέρετε αυτό παράδειγμα για τον αντίκτυπο. Είπατε ότι στην ισπανική περίπτωση η υφαλοκρηπίδα είναι πολύ στενή που σημαίνει ότι οι μικρά σκάφη πρέπει να βγουν ακόμη πιο έξω, σε ανοιχτή θάλασσα. Και άρα ως παραλίευμα μπορούν να έχουν και βαθύ είδη. Αυτό μπορεί να έχει σημαντική στον Ισπανικό στόλο που δεν το λαμβάνεται όμως τελικά υπόψη. Η ανάλυση λοιπόν στοιχεί, ε, στηρίζεται σε ανακριβή στοιχεία για πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένε και της δικής μου. Μου το εξηγήσατε κι εσείς. Απλώς σας επισημαίνω τις αντιφάσεις της μελέτης σας. Και νομίζω ότι οι επιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικές για την Ισπανία. Σας το λέω σε περίπτωση που το αγνοείτε. Επίσης, διασταυρώστε τα στοιχεία αυτά με, το, με τα στοιχεία του πλαισίου συγκέντρωση πληροφοριών. Λέτε στην έκθεση ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην κατηγορία αυτή ένα σημαντικό κράτο, κράτος μέλος δεν έχει χορηγήσει στοιχεία εκφόρτωσης αξίας ή βάρους για καμία από αυτές τις χρονιές, 2008-2011, και τα στοιχεία αυτού του βασικού κράτους μέλους δεν υπάρχουν ούτε για το 2011, ενώ για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη έχουμε ένα ε, ατελή στοιχεία για το 2011. Με όλα αυτά τα στοιχεία κάνατε τις διασταυρώσεις που μας αναφέρατε, με όλα αυτά τα ελλειπή στοιχεία. Μας δώσατε οικονομικά, κοινωνικά στοιχεία, στοιχεία απασχόλησης, αλλά τελικά προς τι όλα αυτά τα δεδομένα, αν τα βασικά κράτη-μέλη ένα δεν έδωσε, άλλο, έδωσε, άλλο κράτος έδωσε ελλειπή στοιχεία, τότε τι μπορείτε να διασταυρώσετε με όλες αυτές τις ελληπείς πληροφορίες. Ξεκινώ λοιπόν από τη βάση ότι είναι ακατάλληλα αυτά τα στοιχεία. Και χθε ακούσαμε το παράδειγμα των καρχαριών που τόσο μας εξέπληξε. Είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η επίπτωση των, ε, της βυθότρατας ε, είναι πολύ διαφορετική από ό,τι η επίπτωση στον υπόλοιπο κόσμο. Το θέμα δεν είναι ότι μας το είπαν μόνο οι, οι αλληλείς, μας το είπαν όλοι οι επιστήμονες που έχουμε, που, που έχουμε καλέσει εδώ. Όλα αυτά δείχνουν ότι στηρίζεστε σε ανακριβή στοιχεία, γιατί και εσείς το αναγνωρίσατε σήμερα είναι πολύ πιθανό όλα αυτά τα στοιχεία να αλλοιώνονται από τις απορρίψεις που έχουν γίνει ε, για τους καρχαρίες. Γιατί επειδή ισχύει μηδενική, μηδενικό τάκ, απαγορεύονται εκφορτώσεις. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς καρχαρίες αλλιεύουν οι μεν και οι δε, μια και μερικοί τους απορρίπτουν. Όλα αυτά που μας λέτε άλλωστε αντιβαίνουν σε αυτά που μας λένε και οι αλείς και οι επιστήμονες. Πώς να στηριχθώ στις δικές σας πληροφορίες. Τι να πω, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Φαίνεται ότι στηριχθήκατε κυρίως στους αλληλευτικούς τόλους ε, που στοχεύουν επί τούτου βαθύβια ήδη. Και παραλείψατε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η παραλίευση. Γιατί δεν έχετε στοιχεία για την παραλίευση. Οπότε α, σας ξέφυγε από την ανάλυση ένα μεγάλο τμήμα του αλληλευτικού στόλου. Και τώρα μετατροπή ε, της βυθότρατας σε παραγαδιάρικο. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα, γιατί λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο το διαφυγόν κέρδος, δηλαδή τα βαθύβια είδη που δεν θα αλλιευθούν στο μέλλον. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη ότι το διαφυγόν κέρδος είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί γενικά μιλούμε για μεικτή αλία δεν αλλιεύεται μόνο ένα είδο, οπότε υπάρχει διαφυγόν κέρδο όχι μόνο εξαιτία μια αλλιεύση βαθύ βιονιδών, αλλά και για τα υπόλοιπα είδη. Δεν θα επισέλθω στο θέμα τη μετατροπή τη βυθότρατα σε παραγαδιάρικο. Χθε αναλύσαμε παρκώ αυτά τα θέματα. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά κοφεύει σε ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Επαναλαμβάνω όμω, τα στοιχεία δεν είναι αρκετά εύγλωτα για μια τόσο σοβαρή δουλειά γιατί αγνοούνται πολύ σημαντικές παράμετροι. Στην περίπτωση του Ισπανικού στόλου τα στοιχεία είναι ανακριβή. Εγώ έχω τα πιο πρόσφατα στοιχεία των αρμόδιων αρχών και παρακαλώ να τα επικαιροποιήσατε, όχι μόνο για την Ισπανία αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ. Μισελ Καντέκ. Σας ευχαριστώ. Επίτηδες το κάνατε. Είναι η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται να σας υποβάλω, κύριε αγαπητή Φουενσάντα. Γιατί το θέμα είναι ήδη πολύ περίπλοκο και λεπτό. Αλλά πραγματικά ή είμαι βλάξ ή τελείως αδαής. Αλλά δεν τα κατάλαβα όλα αυτά. Γι' αυτό και σας ρωτώ, επίτηδες το κάνετε. Δεν νομίζω να το κάνετε επίτηδες. Όχι, εγώ μάλλον είμαι λίγο αρδαής, ε, αλλά ειλικρινά μου διέφυγαν διάφορα κομμάτια. Ένα σωρό προσταφερέσεις εκεί, ε, καταφάσεις και όπως και η συνάδελφος Φράγα, πιστεύω πως αυτή η μελέτη, αυτή ενημέρωση αυτού το της μελέτης αντικτύπου είναι σημαντική, ναι μεν, πολύ σημαντική, αλλά ατελής και έχει πολύ συγκεκριμένο στόχους. Αυτή είναι η εντύπωση που έχω εγώ πάντως. Δεν θέλω να πω τώρα στι λεπτομέρειε, αλλά αν πάρουμε για παράδειγμα το θέμα των ειδών που αλλιεύονται σε μικρές ποσότητες, ξέρετε πολύ καλά για ποια λέω, πάνω από 100 κιλά αναϊχθιόσκαλα. Δεν εμφανίζονται αυτά στην ε, έκθεση αυτή. Ειλικρινά, αυτή η παρουσίαση δεν μου έδωσε κάτι παραπάνω παρά αυτά που ήδη ήξερα και επιπλέον τα περιπλέκει τα πράγματα. Ανησυχώ λοιπόν για το μέλλον και για τις ε, εξελίξεις. Εξάλλου, Κρήτον πριν από λίγο μας έλεγε εισαγωγικά ότι έρονται οι εφηβολίες. Λυπούμε πολύ Κρήτον, αλλά μετά από μια τέτοια παρουσίαση, εγώ έχω πολλές πολλές αμφιβολίες. Λυπάμαι Φουενσέντα, αλλά πολύ ανησυχώ για το τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες γιατί δεν νομίζω πως ε, χρειάζεται σήμερα. Αυτά, Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρωμέβα. Yeah, thank you. Um, Σας ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για το μελέτη αντικτύπου, γιατί νομίζω πως είναι πλήρης και χρειαζόταν. Ζητήσαμε αυτή την αξιολόγηση. Φυσικά υπάρχει το θέμα της έλλειψης ε, ε, δεδομένων, αλλά τα δεδομένα μας τα δίνει το αλληλευτικό τομέας και δεν μας τα δίνει πάντα αυτά που ζητάμε. Επίσης, ε, εμείς όλοι γνωρίζουμε ότι αν, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν δώσει στοιχεία, πλήρη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια ξαφή κατάσταση αντίθετα με τα όσα είπε ο συνάδελφος Καντέκ. Εγώ έμαθα διάφορα πράγματα. Και υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις που θα ήθελα να υποβάλω. Είναι σαφές ότι τα στοχευμένα σκάφη ε, και τα ποσοστά τους είναι πολύ χαμηλά. Τώρα αν είναι 11% ή πάση περιπτώσει είναι κάπου εκεί. Είναι χαμηλό το ποσοστό. Δεν είναι τεράστιος αντίκτυπος που ορισμένοι ισχυρίζονται ότι θα ε, υπάρξει. Δεύτερον, μετατροπή από τις τράτες στα παραγαδιάρικα είναι δυνατή όχι μόνο λόγω του οικονομικού αντικτύπου που μπορεί να έχει, το ανέφερε και η Κομισιόν όσον αφορά την πλήρη κατανάλωση, αλλά και από άπλωση τη σκοπιμότητας. Και φυσικά ο αντίκτυπος αυτή τη δραστηριότητα είναι πολύ χαμηλότερο. μπορεί να το συζητήσουμε το κόστο σα, αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε αργότερα. Και τέλος, τρίτον, υπάρχει κάτι που με απασχολεί και που θα ήθελα να θέσω ερωτήσεις αναφέρατε τα στοιχεία όχι μόνο για τη φύση των ε, στόκ, αλλά και για άλλες ε, υποθέσεις, ας πούμε και για τις περιοχές που πρέπει να κλείσουν. Και με τους εκπροσώπους του κλάδου χτες κάναμε μια συζήτηση είπαν ότι η ΝΕΑΦΚ ήταν το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Στην τελευταία συνεδρίαση η ΝΕΑΦΚ έκλεισε κάποιες ζώνες αλλά όχι όλες αυτές που ζήτησαν ε, οι, οι περιφερειακές, τα περιφερειακά συμβούλια να κλειστούν. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, πώς το αξιολογείτε. Και έπειτα η ΝΕΦΚΑ εξέτασε την προστασία κάποιων ειδών ε, κοραλιών και σπόγγων ε, ε, ψυχρών υδάτων, αλλά δεν έλαβε υπόψη άλλα είδη ευαίσθητων, ευάλωτων για ποιο λόγο επίσης. Για το θέμα των καρχαριών έχω ακόμα κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι μια συγκεκριμένη ερώτηση που έκανα και χθε ε, δεν έλαβα απάντηση. Ίσως εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Υπάρχει κάποια επιστημονική μελέτη που να συγκρίνει τις, ε, τα λιεύματα καρχαριών για τις ε, βυθότρατες και για τα παραγαδιάρικα στην ίδια περιοχή. Έχει γίνει κάποια επιστημονική μελέτη που να δείχνει ότι τόσο τα παραγαδιάρικα όσο και οι βυθότρατες ε, πιάνουν καρχαρίες στην ίδια περιοχή. Ή για να το πω διαφορετικά, ποιες είναι οι περιοχές όπου υπάρχει ε, συγκέντρωση ε, καρχαριών βυθού. Γιατί εκεί όπου ξέρουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση θα έπρεπε να υπάρχει μηδενικό τάκ. Άρα το λογικό είναι αυτέ οι περιοχέ να ήταν κλειστέ. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Υπάρχουν λοιπόν περιοχέ όπου γνωρίζουμε πω υπάρχει συγκέντρωση καρχαριών. Αυτά για την ώρα. Αλλά ίσω να επανέλθω αργότερα. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Πατράου. Ευχαριστώ. Όπως ήδη υπόθηκε, η πρώτη εντύπωση που έχουμε από αυτή την έκθεση αξιολόγηση αντικτύπου είναι όντως ότι είναι πολύ ε, ε, ολοκληρωμένη και περιεκτική και πλήρης. Όμως, με μια πιο προσεκτική ανάγνωση, όπως υπόθηκε και από κάποιους άλλους, <coughs> μας οδηγεί να αμφισβητήσουμε την αξιοπιστία των στοιχείων στα οποία στηρίζονται όλη η μελέτη αν τα στοιχεία που χρησιμεύουν ως βάση για αυτήν εδώ τη μελέτη, τότε και τα αποτελέσματα της ίδιας της μελέτης είναι αμφισβητήσιμα. Η έκθεση εξολόγησης αντικτύπου τονίζει το γεγονός ότι αυτή η μελέτη έχει βασιστεί στα σκάφη που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα VMS, δηλαδή εποπτείας των σκαφών. Και άρα λοιπόν έχουμε συγκεκριμένε ε, ε, σκάφη άνω των 10 μέτρων για το έτος 2011. Έχουμε λοιπόν και ένα μεγάλο κομμάτι μικρών σκαφών που ξεφεύγει από την ε, συγκεκριμένη εξολόγηση που ένα μεγάλο κομμάτι και γνωρίζοντας μάλιστα τη σημασία αυτού του μεριδίου του στόλου για τον στόλο του γενικά τον ευρωπαϊκό πως ε, όταν γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτού του είδους η αλληλεία γίνεται στις ε, υπερπεριφερειακές ε, περιοχές. Άρα λοιπόν εδώ σε αυτή τη μελέτη δεν έχουμε τον αντίκτυπο που θα έχει η πρόταση της Κομισιόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτή την πτυχή γνωρίζουμε επίσης πως τα σκάφη απορρίπτουν ε, τα παραλιεύματα ε, που είναι τα, ε, κάποια βαθύδια είδη και αυτά τα είδη τα οποία μπορεί να υπόκειται σε μηδενικό τάκα γιατί παρότι έχουν αληφθεί δεν υπάρχει καταγραφή των αληφμάτων αυτών. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα σκάφη που καλύπτουν βαθύδια είδη σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό αλλά δεν περιλαμβάνονται στο κομμάτι που αναφέρεται στον ε, στόλο αλληγίες ε, βαθύβιων ειδών, γιατί δεν ξεπερνάνε τα 100 κιλά τα παρελιεύματα. Υπάρχει λοιπόν, για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν, όπως σας εξήγησα, υπάρχει μια κατώτερη εκτίμηση του, ε, του πραγματικού αντικτύπου της πρότασης της Κομισιόν στον στόλο. Και ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην έκθεση, στη μελέτη αυτή, από το πίνακα 23 μέχρι και το 32, Έχουμε τα Κανάρια νησιά ότι είναι 7, η Μαδέρα 2 και οι Αζόρες 2, ενώ είναι 9 τα νησιά των Αζωρών. Και σίγουρα δεν σε κάποιου πίνακε επίση λέει ότι είναι τρία τα νησάκια. Δεν κατάλαβα δύο ή τρία γιατί έχει μια παυλίτσα ανάμεσα. Πάντω σίγουρα δεν λέει εννέα. Άρα λοιπόν δεν είναι πλήρη η τρια γιατι εχει μια παυλιτσα αναμεσα παντω σιγουρα δεν λεει εννεα αρα λοιπον δεν ειναι πληρη εικονα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Άρα όχι μόνο τα στοιχεία είναι ανακριβή, αλλά χάσαμε και μερικά νησιά. Ευχαριστώ πρόεδρε μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που πήραμε ως Επιτροπή είναι ότι επιμικίναμε την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών και ζητήσαμε μια συμπληρωματική έκθεση αντικτύπου και κάναμε μια επιπλέον ακρόαση. Εάν πήραμε αυτή την απόφαση πριν από μερικούς μήνες, όπως είχαν προτείνει τότε, τότε αυτά τα μέλη, εάν δεν είχαμε πάρει αυτή την απόφαση, τότε θα ήταν ε, επιπόλαια η αντιμετώπιση μας. Έχουμε πει ότι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών είναι τον Ιούλιο. Μήπως θα πρέπει, λόγω του πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, πόσο σοβαρέ επιπτώσει θα έχει, μήπως θα πρέπει να παρατείνουμε περαιτέρω την ε, προθεσμία. Η Επιτροπή λέει ότι πολύ λίγα σκάφη θα θυγούν. Άρα, ας το πω απλοϊκά, ε, αν λοιπόν ε, δεν θα θυγούν το 98% των σκαφών, γιατί, γιατί την κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να προστατεύσουμε βεβαίως ε, τα ευάλωτα είδη, τα βυθοπελαγικά και τα ε, ε, θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτός είναι καλός στόχος. Αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να τον επιτύχουμε. Και όταν πρωτεξέτασα το θέμα αυτό και όταν συζήτησα με τον εισηγητή μου είπε «Μα γιατί ενδιαφέρεστε» δεν νομίζω ότι αφορά πολύ τη χώρα σας και νομίζω ότι το είπε καλόπιστα. Αλλά σήμερα έχω πολύ διαφορετική άποψη και ελπίζω να έχει αλλάξει άποψη και ο εισηγητής όταν θα έχει διαβάσει αυτή τη ε, μελέτη αντικτύπου και την παρουσία σήμερα το πρωί. Αν εξετάσουμε τις σελίδες 35 και 44 υπάρχουν μια σειρά διαγράμματα. Υπάρχουν κοιλίδες γύρω-γύρω, γύρω-γύρω στην Ιρλανδία. Θα θυγεί πολύ η Ιρλανδία και μου είπαν ότι η έκθεση αυτή δεν θα είχε καμία επιπτώση για το πράσινο νησί μου. Αλλά τώρα έχουν πρασινίσει οι ακτές του. Και τα διαγράμματα τα λένε όλα πιστεύω. Αν εξετάσετε τη μελέτη επιπτώσεων σελίδα 2, όπου μιλάει για τους βυθοπελαγικούς καρχαρίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, τους πιάνουν οι μηχανότρατες. Αλλά αυτό είναι απόλυτα διαφορετικό από αυτό που μας είπε ο Γερμανός ε, δόκτωρ, ο οποίος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο της Ιρλανδίας, δεν μπορούμε να απορρίπτουμε τις απόψεις τόσο εξεχόντων επιστημόνων που λένε ότι και τα παραγαδιάρικα έχουν επίπτωση και μάλιστα τη μεγαλύτερη στους καρχαρίες. Τι πάμε να κάνουμε λοιπόν τώρα. Και δεν θέλω να τα βάλω με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την ε, εκπόνηση αυτή την έκθεση και αυτούς που εκπροσωπούν την Κομισιόν εδώ σήμερα. Δεν μπορούμε να αγνοούμε, επαναλαμβάνω, τις απόψεις διακεκριμένων και ιδιαίτερα ειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι ενεργά, ενεργά εργάζονται στον τομέα αυτό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα ίδια αυτά, αλλά και τα συμφέροντα της Ένωσης. Δεν μπορεί δεν μπορεί να έχουν και οι δύο ε, αντιδιαμετρικά ε, αντίθετες απόψεις δίκιο και διάβασα στην έκθεση ότι είναι δύσκολο να δούμε τις επιπτώσεις αλλά ας ακούσουμε τους ανθρώπους που ε, δουλεύουν στον τομέα όπως ένας από τους παρουσιαστές χθες μας είπαν ότι το κόστος αυτής της προσπάθειας το κόστος είναι μεγάλο. Αλλάζει συνολικά η δομή του σκάφους από τράτα σε παραγαδιάρικο. Δεν είναι απλό αυτό. Μπορεί να είναι αξιέπαινος ο στόχος. Αλλά δεν τον προσεγγίζουν με τη σωστή προσέγγιση. Αναφέρθηκαν στις εξοικονομήσεις καυσίμων. Μπορεί, μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια θα υπάρχουν. αλλά πρέπει να δούμε και την παρουσίαση του κόστου συνολικά. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν 45-50 ε, παραγάδια που θα πέφτουν. Είναι πολύ ακριβώς αυτή τη στιγμή αυτός ο εξοπλισμός. Είναι πολύ ακριβή η προσπάθεια να αλλιευθούν τα είδη που θα αλλιεύονται με αυτήν την μετατροπή. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά αυτό που κάνουμε. Είτε λίγη η θητεία μας, είτε όχι. Εάν θέλουμε να ε, στοχεύσουμε αυτούς που υπεραλλιεύουν τα βυθοπελαγικά είδη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να κλείσουν κάποιες περιοχές. Ήδη τεράστιες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας και του Βόρειο Ατλαντικού είναι κλειστές για αλληλεία. Και περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας μου. Εντάξει, για μένα είναι πιο σημαντική η χώρα μου, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε στη μέση του Βόρειο-Ανατολικού Ατλαντικού. Αλλά, άρα θα υπάρχουν μεγάλες επιπτώσεις. Στην Ιρλανδία το θαλάσσιο Ινστιτούτο μας έκανε μία αποτύπωση ε, του βυθού των θαλασσών δίνεται εντύπωση ότι επειδή ε, γίνεται αλία στο βυθό, οι τράτες ε, στο βυθό θίγουν και κάνουν ζημιά στο βυθό. Αλλά ξέρετε ότι ε, στο κάτω μέρος του δικτυού υπάρχουν κύλινδροι από καουτσούκ οι οποίοι πηδάνε πάνω από, τις, από το βυθό. Δεν κάνουν αυτή την τεράστια ζημιά που λέγεται στα κοράλια. Όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Ακόμη και αποτίμηση της Κομισιόν αναφέρεται στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας στη σελίδα 11. Οπότε, οπότε, θυμάστε ότι η Επιτροπή μας στην αρχή είπε ότι θα καταργήσουμε τις απορρίψεις, θα τις απαγορεύσουμε και έτσι ως διαμαγείας ε, θα τα λύσουμε όλα. Τελικά αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν ένας συμβασμός. Πιστεύω ότι και για αυτό το θέμα χρειάζεται περισσότερη εξέταση πριν ε, βιαστούμε να αποφασίσουμε. Πρέπει να το σκεφτούμε. Να θυμηθούμε ότι έχουμε δύο βασικές αρχές στη δουλειά μας. Πρέπει να τους επιτύχουμε και τους δύο. Πιστεύω ότι τα παραγαδιάρικα έχουν μεγαλύτερη επίπτωση στα κοράγια από ότι οι τράτες. Αρκούν αυτά πιστεύω. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ. Ο κύριος Αρσένης θέλει να παρέμβει. Μα θα σας άφηνα τελευταίο, αλλά αν θέλετε να μιλήσετε... Μα είχα ζητήσει από την αρχή τον λόγο, λέει ο κύριος Αρσένης. Συνάδελφοι. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κυρίου Καντέκ. Θέλω να ρωτήσω. Τι διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την ε, μελέτη αντικτύπου. Υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Πού είναι αυτά τα στοιχεία. Γιατί εγώ νομίζω ότι η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Ως Επιτροπή εδώ αποφασίζουμε πολύ συχνά τις υποχρεώσεις των χωρών και υπάρχουν ε, αντιπαραθέσεις γιατί ορισμένοι λένε ότι κάποιες χώρες δεν κάνουν όλες τις εκθέσεις που θα έπρεπε. Όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία έχουν τηρηθεί και όλα τα στοιχεία ελήφθησαν υπόψη για την μελέτη αυτή αντικτύπου. Ποια άλλα στοιχεία Πού είναι αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποιος να μου πει ποια στοιχεία δεν λήφθηκαν υπόψη. Για τους καρχαρίες. Εμπιστευόμεθα τα στοιχεία που μας δίνει ο κλάδος. Εμπιστευόμεθα αυτά που μας λέει ο κλάδος ή αυτά που γράφει στα ημερολόγια των πλοίων. Αυτά που μας λένε προφορικά ή αυτά που λένε τα ημερολόγια. Πρέπει να διευκρινίσουμε την κατάσταση. νομικά η αλήθεια, όπως και στις σχέσεις μας, νομικά αυτό που ισχύει είναι το γραπτό. Γιατί αυτό έχει και επιπτώσεις. Ρωτάω την Επιτροπή, γιατί έχουν αφαιρέσει ε, από την πρότασή μου τη λίγκα και τα χέλια. η λίγα και το Μουγκρί, συγγνώμη, είναι χαμηλά τα ποσοστά προσθέμενης αξίας. 1,5% των συνολικών αλλιευμάτων. Γιατί έχουν εξαιρεθεί η Λίγκα και το Μουγκρί. Γιατί έχουν ε, μεγάλη επίπτωση. Ε, μπορείτε να μου κάνετε μια χοντρική εκτίμηση. Για τον κύριο Κάλαχαρ για την Ιρλανδία. Ναι, υπάρχουν πολλά λιμάνια, αλλά το ποσοστό είναι χαμηλό. Παρακαλώ μήπως η Επιτροπή να μας εξετάσει με βάση τα διαγράμματα τα ποσοστά αλευμάτων και αξίας. Για τη Γαλλία. Η Γαλλία, κύριε Καντάκη, ήταν η πρώτη χώρα που μας χορήγησε στοιχεία. Και τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται από την μελέτη είναι τα στοιχεία που μας έδωσε η γαλλική κυβέρνηση. Τέλος για το θέμα της προθεσμίας ε, υποβολής τροπολογιών. Το συζητήσαμε στους συντονιστές. Υπήρξε πλατιά πολιτική συμφωνία και νομίζω ότι ως Επιτροπή σεβόμεθα τις συμφωνίες μας. Ευχαριστώ κύριε Αρσένη. Ε, καταρχάς να καλωσορίσω μια ομάδα επισκεπτών από την Κανταβρία, Κανταβριγία. Ε, συζητάμε θέματα που ενδιαφέρουν πολύ τη χώρα σας. Προσωπικά, να απαντήσω σε μία ερώτηση του κυρίου Αρσένη. Από πού λείπουν στοιχεία. Η κυρία Φράγα έθιξε ένα θέμα σήμερα το πρωί. Οι απορρίψει ε, καρχαριών. Επειδή υπάρχει μηδέν τάκ για τους καρχαρίες, όπως μας είπε η κυρία Καντέλα, μόνο κάποιοι καπετάνοι βάζουν τα στοιχεία αυτά στα ημερολόγια πλοίων για το οποίο ήταν ευγνώμων βεβαίως. Αλλά οι άλλοι πετάνε, απορρίπτουν τους καρχαρίες. Υπάρχουν, λέει ο κ. αυτά τα στοιχεία κάπου. Πού είναι αυτά. Ε, λοιπόν, να αναφέρω το γράμμα της Σαπέσκα. Έχετε μία τράτα 25 μέτρων που αλλιεύει για 10 μέρες. έχει πέντε ε, δραστηριότητες αλίας την ημέρα και πιάνει ένα-δύο κιλά βυθοπελαγικών ειδών που δεν είναι ε, στόχος της, άρα απορρίπτονται. Και επιστρέφουν μετά με 15-20 τόνους ε, αλιευμάτων και σε όλα αυτά ίσως να περιλαμβάνονταν 3-4 κιλά βυθοπελαγικών, Το οποία τα έχουν απορρίψει. Δεν θα πάρουν άδεια για αλληλεία επειδή δεν έπιασαν τέτοιου είδου, επειδή δεν έπιασαν πάνω από 100 κιλά και επειδή τα απορρίπτουν αυτά τα είδη. Δεν έχουμε στοιχεία. Δεν χρειάζεται να τα βάλουν σε μερολόγιο αυτά τα στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Ο κύριο Αρσένη. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι τράτες ε, κάνουν απολογισμό ενώ στα παραγαδιάρικα δεν υπάρχει απολογισμός. Γιατί οι μεν ε, καταγράφουν αυτά οι ειδικοί δεόχοι. Είναι αδύνατο να γίνεται αυτό. Η κυρία Τωμά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Καντέλα και την Επιτροπή γιατί επιτέλους έχουμε στοιχεία. Έχουμε μια έκθεση κοινωνικο-οικονομικής επίπτωσης τουλάχιστον μια εργασία προς αυτήν την κατεύθυνση σημαντική έχει επιτελεστεί. Κρίμα που δεν έγινε στην αρχή της διαδικασίας μια τέτοια μελέτη πριν από ένα χρόνο όταν ε, υπέβαλαν αυτή την πρόταση οι Επίτροποι. Ακόμη και πριν την υποβάλουν οι Επίτροποι θα μπορούσαμε να έχουμε διαπιστώσει ε, αυτές τις ελλείψεις δεδομένων και να τις καλύψουμε. Αλλά τώρα καταλαβαίνω καλύτερα πόσος χρόνος χρειάστηκε γιατί όταν βλέπω τα στοιχεία που μας παρουσιάζουν, χρειάστηκε πολύ ε, ευφυΐα και πολύ ε, ε, μεγάλη προσπάθεια τεχνασμάτων για να συμβιβαστούν τα στοιχεία με τους στόχους της Επιτροπής. Ποια είναι τα θετικά. Πρώτον, προκύπτουν ορισμένες αλήθειες. Όπως είπε και ο Πάντερ Κοπ, αντίθετα με αυτά που μας είχαν πει στην αρχή, δεν αφορά μία-δυο χώρες μόνο. Προφανώς η Μεγάλη κακοί, η Γαλλία και η Ισπανία που πάντα θεωρούνται οι δύο χώρες που επιδιώκουν να αλλιεύσουν τα πάντα, οι χώρες που δεν θέλουν να εφαρμόσουν περιβαλλοντικές ε, διατάξεις. Και όλα αυτά βεβαίως ε, είναι λαθασμένα, θα επανέλθω. Εύκολο λοιπόν να κατηγορούμε και να δαιμονοποιούμε τις δύο χώρες, αλλά όταν μπούμε στις λεπτομέρειες διαπιστώνουμε ότι αφορά όλα τα παράλια του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Και η κυρία Καντέλα έχει σημειωθεί πρόοδος. Είχαμε πει πως θα είναι 1% επίπτωση, τώρα φτάνουμε στο 2%. Άλλη μια προσπάθεια και θα έχουμε τα πραγματικά στοιχεία. Προ την καλή κατεύθυνση λοιπόν πηγαίνουμε. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία. Δεν θα επανέλθω σε αυτά που είπε η κυρία Φράγα. Υπάρχουν πολλά κενά στα στοιχεία αυτά. Αλλά, αλλά, κάτι που είναι πιο σοβαρό. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδα. Όχι μόνο λείπουν στοιχεία, αλλά και η μεθοδολογία είναι ε, αμφισβητούμενη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει αποδεκτή λύση για τις απορρίψεις. Θα γίνεται αποδεκτό ή ανεκτό 7% απορρίψεων, λέγεται τώρα ενώ θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα αλλιεύματα. Όχι μόνο τα αλλιεύματα που εκφορτώνονται, αλλά και τις απορρίψεις ειδών αυτών με μια μεθοδολογία που είναι γνωστή. Πρέπει να εφαρμόσεις μια αναλογία στο σύνολο των δεδομένων. Η απαγόρευση θα έχει και άλλες επιπτώσεις που επίσης δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν ξέρω ποιος το είπε, η κυρία Φράγα ή κάποιος άλλος. Ή η κυρία Πατράου Νέβες. Αν είχαμε λοιπόν στα στοιχεία που έχουμε από το σύστημα VMS για την ανείχνευση της θέσης των σκαφών, θα είχαμε στοιχεία που μπορεί να μην ήταν βέβαια τα τέλεια, αλλά θα ήταν πιο αξιόπιστα. Κάτι άλλο για τη μεθοδολογία. Αυτός ο υπολογισμός της απασχόλησης και το ποσοστό απασχόλησης. Το ποσοστό απασχόλησης είναι 2 έως 4% σε σχέση με τη συνολική απασχόληση. Εγώ ήξερα ότι οι γαλλικές μελέτες πάντα έλεγαν ότι είναι 4 με 6%. Ιδίω για είδη που κατόπιν γίνονται αντικείμενο μεταποίησης. Γιατί όπως είπε ο κύριος Αρσένης, είναι ψάρια που δεν είναι όμορφα. Είναι όμως ε, αντικείμενο μεταποίησης. Και επίσης δεν ελήφθη υπόψη, με συγχωρείτε που μιλάω για θέματα μεθόδου, αλλά ε, ε, είναι η ουσία μιας μεθόδου αντικτύπου, δεν λήφθη υπόψη το φαινόμενο ντόμινο για τις ιχθιόσκαλες ε, που σε μεγάλο βαθμό το κέρδος τους το βγάζουν από τη διαφορετικότητα ε, ειδών. Επίσης δεν λήφθηκε υπόψη η μετακίνηση από ζώνη σε ζώνη. Διότι ε, αν περάσουμε από άλλες περιοχές, τις περιοχές που είναι τα παραγαδιάρικα, εάν χρειαστεί να εισαγάγουμε ποσοστώσεις, επειδή θα υπάρξει πίεση σε κάποια είδη, θα υπάρξει ένα πρόβλημα αποκατάστασης, οπότε κατά συνέπεια ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη προσέγγιση, να μην ε, βασιζόμαστε μόνο στη δύο ποικιλότητα, αλλά και στην ποικιλία των εξοπλισμών. Να προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ζώνες και με τα είδη τον εξοπλισμό των αλλιευτικών. Πιστεύω ότι αν είμαστε λιγότερο δογματικοί και περισσότερη διάθεση συμβιβασμού, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Πιστεύω ότι όντως πρέπει να κλείσουν κάποιες ζώνες. Πιστεύω ότι πρέπει να προσαρμοστεί ο εξοπλισμός στις περιοχές, στις ζώνες και να απαγορευτούν κάποιοι εξοπλισμοί για κάποιες ζώνες. Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο το θέμα, πρέπει να φροντίσουμε για τη διατήρηση κάποιων ειδών. Εγώ προσωπικά είμαι ανοιχτή για οποιαδήποτε συζήτηση που δεν θα βασίζεται σε δογματική προκατάληψη, που δεν θα είναι συνθηματολογικός. Πρέπει να επιδιώξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά να λάβουμε υπόψη και τους οικονομικούς παράγοντες, την απασχόληση και φυσικά και τα οικολογικά θέματα. Και κάτι ακόμη για το κόστος. Για, τις ε, περιφερειακές, για τα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια. Είχαμε μια συνάντηση που ήταν όλα τα συμβούλια παρόντα. Και είπαν όλοι το ίδιο, ότι δεν θεωρούν ότι ακούγεται επαρκώς η φωνή τους και ότι είναι κατά των προτάσεων της Κομισιόν και για το κόστος. Κύριε Ρομέρα, πρέπει να πούμε τα πράγματα από το όνομά τους. Όλα είναι δυνατά, όλες οι μετατροπές καφών είναι δυνατές. Αύριο μπορούμε να ξεκινήσουμε και για το φεγγάρι. Απλώς υπάρχει κόστος. Είναι κόστος. Και ποιος θα το πληρώσει το κόστος. Εδώ μπορούμε να το αποφασίσουμε, δεν θα το πληρώσουμε εμείς. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα με λογικό τρόπο. Όταν παίρνουμε αποφάσεις που έχουν τόσο σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση, πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι και ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τομά. Θα ήθελα να καλωσορίσω και το υπόλοιπο των επισκεπτών από την Καντάβρια. Καλώς ήρθατε συνεχίζουν, συνεχίζονται πολυάριθμοι, πολυπληθέστατοι αυτή η ομάδα των επισκεπτών από την Καταβρία. Η Σαμπέλα Λεβίν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις προσπάθειες ε, που έκανε προκειμένου να εκπονήσει την συμπληρωματική μελέτη επιπτώσεων επί της προηγούμενης μελέτης και της προπροηγούμενης μελέτης επιπτώσεων ε, πολύ συζητημένο το θέμα. Συμφωνώ ότι πολλοί άριθμα είναι και τα στοιχεία και οι αριθμοί και σίγουρα ε, η έλλειψη των στοιχείων δεν βαρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα κράτη-μέλη υπεύθυνα για μη υποβολή δεδομένων και άλλωστε και δεν είναι και πρώτη φορά. Ε, πρόσφατα, στα στοιχεία και τις επιχορηγήσεις καυσίμων, μερικές χώρες δεν δίνουν στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμων. Οπότε, πώς να κάνει την ανάλυση της Επιτροπή εφόσον δεν της χορηγούνται τα απαραίτητα στοιχεία. Διαπίστωσα από την παρουσίασή σας ότι 1116 αλληλευτικά είδη ε, καλύπτονται, είναι βαθύβια δηλαδή. Και όταν μιλούμε για την έλλειψη δεδομένων και το επίπεδο της γνώσης, Έχω μία γενική ερώτηση. Τι γνώσεις έχουμε για αυτά τα 1116 ελληνικά είδη των βαθαίων υδάτων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζονται από αυτή την αλληλευτική προσπάθεια και 25 μόνο από αυτά τα 1116 είδη υπόκειται σε κάποια όρια. Και τα τρία βασικά είδη που έλεξα εγώ από τις στάσεις του Διεθνού Συμβουλίου Εξερεύησης των Θαλασσών ε, πιστεύω ότι μας ε, ε, δείχνουν την πραγματικότητα. δεν είναι γνωστή για το μαύρο σπαθόψαρο η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Για τη μουρούνα επίσης δεν είναι γνωστές οι αποδόσεις, οι μέγιστες αποδόσεις. Για τη λίγκα έχουμε ορίμανση σε μήκος 75 εκατοστά με βάση την ISIS σημαντικό τμήμα των αλλιευμάτων αφορούν μη όριμο ψάρι. Για το γρεναδιέρο των βράχων ζει 70 χρόνια. Η χρησιμότητα των ψαριών και η βιομάζα για τα, τα ίδια αυτά είναι άγνωστες. Παρακαλώ λοιπόν θερμά. Μην βγάζετε το μεγεθυντικό φακό και δηλίστε τον κόνοπα για κάθε μικρό τμήμα ε, της του κάθε αλληλευτικού στόλου και τον αντίκτυπο που έχει η πρόταση αυτή για τους στόλους αυτούς ενώ ταυτόχρονα εθελοτυφλούμε, θα πρέπει να, λάβουμε, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και για το μέλλον των ευρωπαϊκών θαλασσών και να προστατεύσουμε αυτή την βιοπικιλότητα, να τη διαφυλάξουμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και για τις επερχόμενες γενναίες. Γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι καταστρέφουμε στους βυθούς των θαλασσών. Ελάχιστες είναι οι γνώσεις και τα στοιχεία που έχουμε ακόμη και για τα τρία βασικότερα εμπορικά είδη, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα ελευτικά αποθέματα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και μία ακόμη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνατε αυτή τη μελέτη επιπτώσεων επί του αντικτύπου του αντικτύπου. Οπότε, ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα, επιφέρατε, που θα στην πρότασή σας μετά από την ενημέρωση των στοιχείων. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές μετά από τι τελευταίε αυτέ μελέτε επιπτώσεων. Τέσσερι ακόμα μιλητέ έχω ζητήσει το λόγο. Θα ολοκληρώσω. Ε, πρέπει να κλείσω τον κατάλογο γιατί έχουμε και άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Κυρία Ρόντουστ. Ε, ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη, γιατί ήδη υπόθηκαν πολλά. Καταρχάς, ευχαριστώ την Κομισιόν και νομίζω ότι έχουμε ένα σημαντικό έγγραφο που προσθέτει στη μεγάλη συζήτησή μας. Το χρειαζόμασταν. Θα ήθελα να πω δύο λόγια στον συνάδελφο Καντέκ. Είμαι πεισμένη ότι η Κομισιόν αξιοποίησε όλα τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της. Δεν είναι δυνατόν να τους επικρίνουμε εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Παρακαλώ να επικρίνουμε εκείνους οι οποίοι δεν χορηγούν αυτά τα στοιχεία. Συμφωνούμε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές μεγάλου βάθους, στις θάλασσές μας. Θέλω να το τονίσω. Με συγχωρείτε που ε, στρέφουμε κατά συγκεκριμένου ατόμου κάνω προσωπική επίθεση, αλλά δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς αυτής, αυτός. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, έχουμε αφιερώσει πολύ χρόνο, έχουμε κάνει δύο μεγάλες έκτασεις ακροάσεις, έχουμε διάφορα κείμενα. Ήρθε η ώρα επιτέλους να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να αποφασίσουμε μεταξύ μας πώς θα αποφασίσουμε. Αυτό το σπαγκάτο από τη μία μεριά οι ανησυχίες των επιστήμων από την ε, πρώτη ακρόαση να τονίζονται τόσο πολύ και από την άλλη πλευρά να λαμβάνεται τόσο ε, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα συμφέροντα του κλάδου είναι ένας δύσκολος συμβασμός αλλά εάν δεν έχουμε παρκή στοιχεία και εάν ξέρουμε ότι θα μπορούσαν να ήταν τρομερές επιπτώσεις ε, από την ε, ανεπίστρεπτη καταστροφή των βυθών. Αν ξέρουμε ότι ε, πιάνουμε ψάρια που μπορούν να ζήσουν 150 χρόνια, τότε έχω πρόβλημα εγώ. Και αν πούμε, οκ, okay, να βάλουμε παραγαδιάρικα. Αν μας λέτε ότι αυτό είναι πολύ ακριβό και είναι ακριβή η αλλαγή του εξοπλισμού και ακριβή η κατάρτιση των αλλιέων, η επανεκπαίδευση, ε, τότε να σταματήσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Αν θέλουμε παραγαδιάρικα. Για μένα το να συνεχίσουμε αυτά ε, με τις μηχανότρατες βυθού δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Πρέπει να είμαι σαφής. Χάτσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία με κάτι που θα είναι λογικό και εύχριστο να βρούμε μία χρυσή τομή μεταξύ των απόψεων ε, του κυρίου Γκάλαχαρ και άλλων και της κυρίας Λέβεν και τις ανάγκες δηλαδή που είναι κοινή για όλους να έχουμε ε, υγιείς ελευτικούς πόρους ε, και καλά διατηρημένο βυθό και θαλάσσια οικοσυστήματα. Χθες ένας εμπειρογνώμονας επισήμανε ότι ε, αυτοί που θα βγουν περισσότερο κερδισμένοι από επιτυχή διατήρηση των ελευτικών πόρων είναι οι Ο κύριος Πάρκα, δεν κάνω λάθος, είπε χθε ότι οι βυθότρατες δεν ε, χρησιμοποιούν και θελώς τα ακριβά ε, ελευτικά εργαλεία τους και δεν τα φθήρουν επειδή το επιθυμούν ούτε θέλουν να καταστρέφουν ευαίσθητους βυθούς που περιέχουν κοράλια, σπόγκους ή άλλα οικοσυστήματα. Πραγματικά κατακλειστήκαμε με στοιχεία σε αυτές τις πολλαπλές μελέτες επιπτώσεων. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει δεν είναι να μας πει η Επιτροπή με να ανησυχείτε μόνο το 2% του στόλου θα επηρεαστεί από την πρόταση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιο είναι αυτό το 2% και ποια είναι η εμφάνισή τους, η συγκέντρωσή τους σε συγκεκριμένες αλληλευτικές κοινότητες. Εγώ εκπροσωπώ εδώ ένα αλληλευτικό έθνος στη Σκοτία και όπως είπε ο κύριος Πάρκ, δεν θέλουμε ανεπιθύμητες συνέπειες ε, και ιδιαίτερα αν ε, αποδειχθεί ότι το σύνολο των σκαφών της σκοτικής αυτής κοινότητας θα επηρεαστεί και αν ε, ήταν υποχρεωτική μετατροπή από βυθότρατε σε παραγαδιάρικα, αυτό θα οδηγούσε σε καταστροφή της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή αυτή. Και να τους πούμε μην ανησυχείτε, ανήκετε μόνο στο 2% της ευρωπαϊκής, ε, του ευρωπαϊκού στόλου που πειράζεται από την πρόταση, δεν νομίζω ότι θα τους παρηγορήσουμε αν οι άνθρωποι καταστραφούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφήνεια και διευκρινήσεις για τον ακριβή αντίκτυπο σε συγκεκριμένα τμήματα του στόλου, αν τελικά ευοδοθεί αυτή η πρόταση. Γιατί δεν μας αρκούν κάποιες καθησυχάσεις ότι είναι δυνατή μετατροπή βυθότρατα σε παραγαδιάρικο. Ε, είπατε ότι θα χρειαστεί 300.000 ευρώ ανασκάφο με βάση τα σημερινά στοιχεία. Ποιο θα πληρώσει όμω αυτά και ποιο θα είναι το κόστος ε, του παροπλισμού αυτού του πλοίου. Για πόσο καιρό θα χρειαστεί ε, να γίνει μετατροπή, πόσου μήνε. τι γίνεται με το δευτικό κέρδος, όσο διαρκεί αυτή η μετατροπή του σκάφου, Όλα αυτά θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν σε μια μελέτη οικονομικών επιπτώσεων που θα πρέπει να συνοδεύει τις προηγούμενες. Οι συνέπειες λοιπόν, επιθυμητές, ανεπιθύμητες, θα πρέπει να δοθούν όχι μόνο με γενικούς ε, και ενοποιημένου ε, πίνακες όπως είδαμε και στη μεταρρυθμίση ΚΑΠ, αλλά συγκεκριμένους πίνακες για τον αντίκτυπο σε συγκεκριμένες αλληλευτικές κοινότητες και μικρές όπως είναι η Δυτική Σκοτία, αλλά και εκεί που έχουμε τις μεγάλες ε, κουκίδες, Βορειοανατολική Σκοτία, Σέτλαντ, γιατί εδώ και χρόνια έχουμε πληγεί από ατυχείς εμπειρίες εφαρμογής της κοινής ελευτικής πολιτικής και είχαμε πραγματικά ύφεση της οικονομικής δραστηριότητας εξαιτία της ρύθμισης. μη μου λέτε λοιπόν να μην ανησυχώ επειδή μόνο το 2% του, στόχου, του στόλου επηρεάζεται από την πρόταση. Πείτε μας ακριβώς ποιες θα είναι οι συνέπειες στη σκοτία. Τότε μόνο θα μπορέσω να εξετάσω τον κανονισμό και να αποφανθώ αν αξίζει να εγκριθεί ή μήπως ε, θα πρέπει να θετήσουμε άλλα μέτρα για να υλοποιήσουμε τους στόχους της διατήρησης των ε, ελευτικών πόρων. Ο κύριος Μιλάνα. Κοιτάξτε, αν ε, είχαμε προσέξει τόσο πολύ όταν γκρίναμε και το κανονισμό για τη Μεσόγειο, μάλλον δεν θα τον είχαμε γκρίνει ποτέ. Μάλιστα, αν είχαμε προσέξει τόσο πολύ, σημερινή η ψηφοφορία για τη δική μου έκθεση θα έπρεπε να ψηφιστεί ακόμη περισσότερο. Γιατί θα έπρεπε να είχαμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο κοινωνικός αντίκτυπος ορισμένων κανόνων να μην ληφθεί υπόψη. Μα ξυπνήστε φίλοι μου, εδώ είμαστε μια κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το τέχνασμα της αναβολής για να μην κάνουμε κάτι έχουμε ε, που και που το δικαίωμα να λέμε, και το καθήκον μάλλον να λέμε όχι στην Επιτροπή, αν δεν είναι εντάξει τα πράγματα. Γιατί η αίσθηση που εγώ έχω είναι ότι έχουμε φτιάξει ένα θεατράκι όπου τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε δεν έχουν στόχο να συζητήσουμε από της ουσίας, αλλά να μην συζητήσουμε σε αυτή τη θητεία, αυτή, τη, το, νομοθέτημα. Γι' αυτό και δεν λέω τίποτα επί της ουσίας. Λέω απλά ότι έχουμε ορίσει μια ημερομηνία προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και συμβουλεύω τον συντονιστή μου να μην αλλάξει αυτή την ημερομηνία. Εγώ στο δικό μου αυτό συμβουλεύω τώρα αν γίνει τέτοια πρόταση πούμε, για αναβολή, αλλά το σημείο κλειδί αυτή τη υπόθεση είναι ότι εμεί στην Επιτροπή την Κοινοβουλευτική έχουμε το καθήκον να απαντήσουμε σε μια πρόταση τη Κομισιόν που είχε όλο το χρόνο, είχαμε όλο το χρόνο γιατί χωνέψουμε και με το παραπάνω και σήμερα όσοι δεν συμφωνούν ας καταψηφίσουν. Πρέπει να καταψηφίσουν. Δεν πρέπει να καθυστερεί. Να πει όχι, απορρίπτω την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά όχι να προσπαθεί να αλλάξει τη φύση της, τη δομή της. Τώρα, έπειτα, αν υπάρξει πλειοψηφία προχωράμε, ναι, λέει ναι, αν όχι, όχι. Γιατί, τι θα κάνουμε, τους ηθοποιούς σε μια κομμαδία, δεν ε, είμαστε εκπρόσωποι των, της πραγματικότητας στην Ευρώπη. Η κυρία Γκαρσία Χιάρο. Καταρχήν, θα ήθελα να καλωσορίσω τους συμπατριώτες μου από την Ισπανία, από την Κατάβρια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ήρθαν στην Επιτροπή και παρακολουθούν τις συζητήσεις μας. Ε, φαντάζομαι ότι θα διαφωνήσουμε στο σημείο αυτό. Δεν θα αναλύσω τη γνώμη μου. Αν ήταν να μιλήσουμε για μουσικά κομμάτια, δεν θα έλεγα οπερέτα, θα έλεγα σαρσουέλα, που είναι υποκατηγορία. Είναι τόσο αφιλεγόμενο αυτό το θέμα και φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο πόλοι. Στον ένα πόλο είναι αυτοί που λένε ότι δεν έχουμε όλα τα στοιχεία ή είναι ανακριβή ή είναι συγκεχημένα ή δεν χορηγούνται ή δεν έχουμε δηλώσεις ε, για τον αντίκτυπο και, στον, και ταυτόχρονα έχουμε περικοπές, θα γίνουν ζημίες, θα πρέπει να δοθούν επιχορηγήσεις και υπάρχει και ο άλλος πόλος, υπάρχει και το πρίσμα το, της παράκτητης αλίας, των μικρών αλληλίων, που ασχολείται με βιώσιμη αλεία που δεν χρησιμοποιούν μεγάλα σκάφη, δεν ρηπαίνουν το περιβάλλον, δεν έχουν μεγάλα δίχτυα ε, σειρώμενα που καταστρέφουν τους βυθούς. Ακούσαμε χθες ε, εκπροσώπους τους, ε, δημιουργούν πάνω από 14.000 θέσεις εργασίας άμεσα και είναι αυτοί που έχουν, ε, τους, έχει ξεχάσει η κοινή αλληλευτική πολιτική γιατί δυστυχώς ε, είναι μεγάλη λησμονημένη γιατί δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε μέτρα και υπέρ αυτών των αλλιών μικρής κλίμακας. Έχουμε εδώ 40 πλοία λέμε ή 164 συνολικά. Μας απασχολεί αυτό το στοιχείο, μας προβληματίζει. Και με κάθε σεβασμό θα έλεγα να σας, θα σας έλεγα ότι δεν θα πρέπει να ανησυχούμε περισσότερο για αυτούς από ότι για τους μικρούς ελίες, γιατί εκεί ούτως ή άλλως οι μεγάλοι ελίες έχουν πολύ περισσότερη οικονομική άνεση να κάνουν επενδύσεις και να προσαρμοστούν στις ανάγκες της βιώσιμης ελίας. Τις προάλλες η κυρία Ρόντους είπε ότι στην Γερμανία δεν επιδοτούνται συγκεκριμένοι κλάδοι, ούτε στη δική μου πατρίδα. Πολλοί τομείς και πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί ανεξάρτητοι ελεύθεροι επαγγελματίες ξεκινούν ε, τη δουλειά τους, ε, υποθηκεύουν τη ζωή τους, την προσωπική, την, οικογενειακή και δεν πάνε καλά. Ούτε πίστευαν ότι εξαιτία μια συγκεκριμένης ε, νομισματικής πολιτικής ή δημοσιονομικής πολιτικής ε, για την οποία δεν έχουν αυτή καμία ευθύνη θα υποστούν μειώσει μισθών ή θα τους απολύσουν ή θα τους κάνουν έξωση. Και μάλιστα όταν μιλούμε για ένα πολύ σημαντικό από οικονομική άποψη κράτο όπως είναι η Αλία, ε, δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε θέσεις που ευνοούν κάποιους ε, και αδικούν άλλους. Αυτό είναι το δίλημα. Αν υπάρχουν στοιχεία τα κάτι μέλη υποχρεούνται να τα χορηγήσουν. Αυτό ανέκαθεν το ζητούμε. Το είπα και στην ε, κοινή οργάνωση αγοράς, ε, στα, στη Γεωργία, το είπα και αλλού. Γιατί αν θέλουμε ε, θάλασσες και θαλάσσια οικοσυστήματα και στην Ευρώπη και αλλού, με σωστές προδιαγραφές, θέλουμε και ε, σκάφη όταν αλλιεύουν να τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές. Να μην εφαρμόζουμε αυστηρές προϋποθέσεις ε, στην Ευρώπη και να είμαστε υπερβολικά χαλαροί και ποιικοί για το ότι γίνεται στις τρίτες χώρες. Γιατί ο καθένας εκπροσωπεί το εκλογικό του σώμα. Δεν είμαστε και αθώς περιστερές. Ε, φυσικά θέλουμε ε, λογική και βιώσιμη αλληλεία και ξέρουμε ότι ε, ε όταν ε, χρησιμοποιούν μικρά δίκτυα είναι καλύτεροι, όταν χρησιμοποιούν καμάκι δεν μπορούν να αλλιεύσουν παντού εξαρτάται και από τις αλληλευτικές ζώνες. Ε, φαίνεται, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, ότι δίνουμε υπερβολική έμφαση σε ορισμένα θέματα. Γιατί η δήλωση επιπτώσεων ήρθε την Παρασκευή και μάλιστα μόνο στα αγγλικά αυτή η μελέτη των επιπτώσεων. Και δεν είναι ότι δεν έχουμε μεταφραστές, αλλά πιστεύω α, ότι δικαιούμαστε στους Ισπανοί να έχουμε ε, την ισπανική μετάφραση. Νομίζω ότι όλες οι μητρικές γλώσσες ε, που αυτές που αναγνωρίζουν στην Ενώση θα πρέπει να εξασφαλίζουν μεταφράσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχω την εφαλιότητα, ούτε την ηρεμία ε, για να αποφανθώ ε, έχοντας δημιουργήσει εμπεριστατωμένη άποψη. Τι θέση βρίσκομαι. Σε αυτή την μεταβατική περίοδο που θα πρέπει να την περάσουμε όλοι, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε να μην πλήξουμε οικονομικά τον κλάδο, για να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται αυτή η μετάβαση, ούτε να θυγούν θέσει απασχόληση. Αν βρούμε λοιπόν αυτή τη χρυσή τομή, μακάρι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε όλα τα μέσα. Και όταν λέω όλα τα μέσα εννοώ όλα και από όλους. Δεν να κατηγορώ μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί φαίνεται ότι πολύ βεβαιασμένα λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις, άρον-άρον, ε, και κάπως επιπόλαια σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την απασχόληση, συγκεκριμένες περιφέρειες, αλληλευτικές κοινότητες, ε, τους ψαράδες τους, τις οικογένειές τους και φυσικά με απασχολεί και το περιβαλλοντικό ε, σκέλος. Αλλά δεν έχουμε κανένα θαυματουργό ε, δίχτυ, κανένα θαυματουργό αλληλευτικό εργαλείο δεν μας λένε κάτι τέτοιο τα στοιχεία. Οπότε από τη στιγμή που δεν μας λένε κάτι τέτοιο τα στοιχεία, οι κανόνες θα πρέπει να είναι σαφείς και να δούμε ποια ηλεκτρικά είδη και πού θα προσέξουμε και θα απαγορεύσουμε. Αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Κανένας δεν μας υποχρεώνει. Κανένας κανονισμός δεν μας υποχρεώνει να λάβουμε απόφαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν μας πιέζει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο και δικαιούται να διαμορφώσει εμπεριστατωμένη γνώμη. Εγώ δεν έχω ακόμη τέτοια γνώμη. Για... Σε, σε τέτοια περίπτωση προτιμώ τον προηγούμενο κανονισμό που λειτουργεί εδώ και χρόνια. Μερικοί από τη βιομηχανική ελεία με κατακρίνουν ότι δεν είμαι και πολύ ευχάριστος άνθρωπος, αλλά προσοχή να μην διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα των αλληλευτικών ειδών των βαθαίων υδάτων. Υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσει για την Ισπανία από την πρόταση. Και δεν μιλάω μόνο για την γαστρονομική άποψη. Είναι θέμα πολιτισμικό. Έχουμε ολόκληρες περιφέρειες που ζουν από αυτό και έχουμε πολύ κόσμο που πηγαίνει στις περιοχές αυτές και απολαμβάνει όλες αυτές τις ε, παραδόσεις και την ισπανική γραστρονομία. Αν ένα, κείμενο, ένα λευτικό είδος ε, βρίσκεται σε κίνδυνο θα πρέπει να λάβουμε ε, τα απαραίτητα μέτρα συγκυριακά ή περιπτωσιολογικά όπως έγινε και με τον τόνο. Το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Δεν είναι ούτε θέμα προσωπικών απόψεων, ούτε αν θέλουμε να γινόμαστε αρεστοί όχι. Θέλουμε όλα τα στοιχεία από όλου. Μόνο έτσι θα διαμορφώσουμε τεκμηριωμένη άποψη. Για να είναι και σωστή και ισορροπημένη. Γιατί φοβάμαι ότι ήδη βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Και ναι, μεν υποστηρίξαμε κάποιες προτάσεις ε, ε, γιατί ανήκουμε σε μια ομάδα, θα σταματήσουμε να υποστηρίζουμε μερικές γιατί είμαστε αφοσιωμένοι και στη, στη συμφέροντα της πατρίδας μας. Το λέω καθαρά και εξάστερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στην κυρία Καντέλα και σας παρακαλώ, σας δίνω πέντε λεπτά, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά παρακαλώ να απαντήσετε σε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι. Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Σε σχέση με την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που σχολιάστηκε πολύ. Να σας πω το εξής, ε, Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής. Εμείς ε, μα, ε, μας έδωσε θάρρος αυτή η προσπάθεια. Ξέρουμε τις δυσκολίες που έχουν σήμερα τα κράτη-μέλη στη συλλογή στοιχείων. Όλοι έχουν δυσκολίες δημοσιονομικές κτλ και το πλαίσιο συλλογής δεδομένων υποχρεώνει τα κρατημέλη να ομαδοποιούν τα δεδομένα και να τα επεξεργάζονται. Και αυτό παίρνει χρόνο και χρήμα. Αλλά αυτό που κερδίσαμε με αυτή την ανάλυση είναι ότι ζητήσαμε τα κατέργαστα υλικά. Ζητήσαμε πολύ βασικά στοιχεία για τα αλευτικά ταξίδια ανασκάφη και εμείς τα ομιδοποιήσαμε εμείς ίδιοι. Γι' αυτό ήταν κάτι που ήταν πολύ θετικό το γεγονός, δηλαδή ότι πήραμε ένα έτος πλήρων στοιχείων από όλους που δεν που, που ενδιαφέρονται την πρόταση. Τα στοιχεία είναι αυτά που υπάρχουν όντως και πιστεύω πως είναι, έγινε μια αναφορά ε, για τα, στα μικρότερα σκάφη από διάφορους ε, βουλευτές. Τα μικρότερα σκάφη δεν χρειάζεται να φέρουν το VMS ε, ούτε και γραπτό ημερολόγιο πλοίο. Και αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν με την προϋπόθεση ότι τα μικρότερα σκάφη αναλογικά θα ληφθούν υπόψη. Άρα λοιπόν έχουμε συλλογή στοιχείων, κάποια τα, συλλέγουν και τα ομαδοποιούν. Αλλά δεν έχουμε μεμονωμένα στοιχεία γιατί θα ήταν πολύ μεγάλο βάρος για τους μικρούς αλληλείς να, να, είναι αναγκασμένοι να αναφέρουν με τον ίδιο τρόπο που αναφέρουν ε, τα μεγάλα σκάφη της βιομηχανικής αλληλείας. Είναι μια αποδεκτή αρχή, είναι τμήμα της δομής της κοινή ελεκτική πολιτικής και είναι ένα τίμημα το οποίο το έχουμε δεχτεί ε, προς το συμφέρον του αλευτικού τομέα και των μικρών ε, ε, κοινοτήτων που λειτουργούν. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι που μπορέσαμε να τα συγκεντρώσουμε και να σας τα παρουσιάσουμε. Και ένα μικρό κομμάτι ε, το οποίο επίσης αναφέρεται σε πολλές ερωτήσεις, είναι τα 100 κιλά. Είπατε, υπόθηκε μάλλον ότι ο αντίκτυπος της πρότασης στα άτομα τα οποία απορρίπτουν σήμερα δεν περιγράφεται εδώ. Ο αντίκτυπος της πρότασης για τους ε, ανθρώπους που απορρίπτουν είναι μηδενικό. Γιατί αν δεν απορρίπτουν αυτά τα, αυτά τα ε, ψάρια δεν κερδίζουν τίποτα. Είτε, είτε αλλιεύουν είτε όχι δεν έχει νόημα. Ε, γιατί δεν τα εκφορτώνουν. Αν στο μέλλον χρειαστεί να εκφορτώσουν ε, τις, ε, τα λιεύματά του υπό την απαγόρευση απόρριψης, τότε θα πρέπει να δούμε αν έχουν ποσόστοση ή όχι. Και αυτό θα ορίσει το βάρος και όχι αυτή την πρόταση. Εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν άδεια σήμερα, δεν χρειάζεται να έχουν και αύριο απαραίτητο άδεια η επιστολή φαίνεται να έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση στις αλληλευτικές ζώνες. Εάν δεν έχουν αποσώστοση στο μέλλον για να εκφορτώσουν αυτά που αλλιεύουν, θα χρειαστεί να λειτουργούν στις ίδιες περιοχές όπου λειτουργούν τώρα και θα πρέπει να εκφορτώνουν το αλλιευμά τους, αλλά πιθανότατα δεν θα τους επιτρέπεται να το πουλήσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με την πρόταση τούτη. Η πρόταση αυτή δεν σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι που τώρα απορρίπτουν δεν θα μπορούν να αλλιεύουν. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την άδεια στην ανοιχτή θάλασσα ή όχι. Ε, δεν σημαίνει ε, ότι δεν μπορείς να, ψηφ... να αλλιεύσεις μερλούκιο ή άλλα είδη. Δεν μπορείς όμως να πουλήσεις τα παραλιεύματα ε, βαθύβιων ειδών που μπορεί να έχεις. Ο οικονομικός αντίκτυπος της πρότασης αυτής σε αυτούς όλους είναι μηδενικός. Ευχαρίστως να σας το εξηγήσω άλλες 100 φορές αν θέλετε, Πρόεδρε. Έλαβα και άλλη μια ερώτηση για το κλείσιμο διαφόρων ληφτικών ζωνών. Η ΝΕΑΦΚ δεν έχει πάντοτε καταφέρει να συμφωνήσει για τα όρια των ε, περιορισμένων ζωνών. Έχουν, ε, θέλουν να διευρύνουν την περιοχή και πρέπει να δούμε τι θα γίνει στην ετήσια ε, συνεδρίαση. Χρειάζεται συνένεση όλων των συμβαλωμένων μερών. Ρωσία είναι μέσα, Ισλανδία, Ενίση Φερόες, Ένωση. Έχουν γίνει απόπειρε για να διευρυνθεί παλιότερα δεν εξευρέθη συνένεση. Για τον κύριο Γκάλαχερ και τον κύριο Χάτσον, αλλά και τον κύριο Αρσένη, που θελήσατε να, να, να, να αποσαφηνίσουμε την κατάσταση με τις ε, τελείες. Είδατε η Ιρλανδία και η Ηνωμένο Βασίλειο αλλιεύουν ε, το Λίγκα ή η μουρουνα Είναι και το κύριο αλλιεύμα. Άρα λοιπόν οι εκφορτώσεις είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει όμως να δούμε τι σημαίνουν οι εκφορτώσεις αυτές για την αξία ολόκληρης της περιφέρειας. Και σε αυτή την περίπτωση είναι κάτω από το 3%. Αυτές οι αλλιεύσεις λοιπόν μουρούνας πληρώνουν για απασχόληση, για θέσεις απασχόλησης που είναι το 3% της τοπικής οικονομίας. Ναι, υπάρχουν ε, τελείες, αλλά όπως είπε και ο κύριος Αρσένης θα πρέπει να δούμε ε, τα νούμερα, να δούμε δηλαδή τι αντιπροσωπεύει αυτό για την οικονομία της περιοχής κάθε φορά. Well, Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα εγώ να κάνω προβλέψεις με βάση τα στοιχεία, αλλά είναι αλήθεια αυτό που είπατε κύριε Αρσένη, ότι η λίγα η Μουρούνα και οι, και Γαρίδες είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συνολιακών ελιγμάτων και θα υπάρξει συνέπεια, αλλά δεν μπορώ να την ορίσω ακριβώς, οπότε δεν θα εκφραστώ. Τέλος, ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω για την ερώτηση της κυρίας Λάβιν για το τι θα γίνει με τον αριθμό των ειδών που απαριθμώνται εδώ. Έχει παραθέσει σωστά τις συμβουλές του, την, την, της ISIS εδώ έχει εφαρμοστεί μια νέα προσέγγιση στις τελευταίες ε, υποδείξεις. Δεν ξέραμε όμως ακριβώς την ε, βιομάζα, τη βιωσιμότητα, η ISIS θέλησε να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ε, δυνατότητες αναλυτικής αξιολόγησης και έφτασαν αρκετά κοντά σε πλήρη αναλυτική αξιολόγηση για τον ε, γρεναδιέρο των βράχων, ενώ σχεδόν το ίδιο έγινε και με το μαύρο σπαθόψαρο. Εμείς στην Κομισιόν θεωρούμε πως γνωρίζουμε αρκετά για αυτά τα δύο είδη για να ξέρουμε ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση ακόμα και δεν έχουμε απόλυτα ακριβή στοιχεία. Και τα υπόλοιπα είδη όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι είναι σε περιορισμένη κατάσταση τα στοιχεία που έχουμε και για τα υπόλοιπα εκατοντάδες είδη δεν έχουμε καμία απολύτως συμβουλή που είναι τα παραλιεύματα. Για να απαντήσω αν θέλουμε να αν προτιθέμεθα να αλλάξουμε την πρόταση τώρα. Μπορώ μόνο να πω ότι το έγγραφο που έχετε ενώπιόν σας ε, σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνει τις αρχικές, τα αρχικά ευρήματα. Στην αρχική αξιολόγηση αντικτύπου είπαμε ότι αν δούμε το σύνολο του όγκου της αλληλείας βαθύ βιονιδών μόνο ένα μικρό ποσοστό της οικονομίας των το, του αλληλευτικού στόλου αντιπροσωπεύουν και είπαμε ότι ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί τοπικά να υπάρχουν ε, ε, συγκεντρωμένες ε, επιπτώσεις και αυτό ακριβώς μας έδειξε και αυτή η μελέτη η οποία μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες και ακρίβεια. Πάντως επιβεβαιώνονται τα αρχικά μας ευρήματα και πορίσματα. Τα στοιχεία λοιπόν σας τα παρουσιάσαμε και μπορούμε και να αποσαφηνίσουμε οποιαδήποτε άλλη πτυχή επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε. Κύριε Αρσένη, δύο λεπτά maximum αν μπορείτε. Νομίζω πως ήταν πάρα πολύ καλή η συζήτηση με πολλές εντάσεις κάποιες ε, στιγμές, αλλά αυτό είναι καλό στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ε, να έχει ο καθένας τη γνώμη του και να την υποστηρίζει. Είναι σαφές ότι όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, όλα τα στοιχεία που, έχουν, που, υπάρχουν έχουν χρησιμοποιηθεί και ότι Όποια στοιχεία, οποιαδήποτε στοιχεία χρησιμοποιούνται ε, επί τη βάση των ημερολογίων των πλοίων και των επισήμων δηλώσεων του κλάδου και για τους καρχαρίες, ας πούμε για την περίπτωση της Ιρλανδίας και των βορειότερων θαλασσών, τα βασικά τα λεύματα είναι μικρά, πολύ μικρά. Ε, αυτό που προτείνω εγώ, επί τη βάση ε, επιστημονικών ε, στοιχείων, θεωρείται ότι είναι αποδεκτό από την Επιτροπή και αυτό σε σχέση και με τον Μουγκρή, Σημαίνει δηλαδή ότι τελικά αυτή η πρόταση δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση. Αυτά τα πράγματα λοιπόν νομίζω πλέον έχουν αποσαφενιστεί μετά από αυτή τη συζήτηση. Και το επόμενο ραντεβού θα πρέπει να είναι στις 8 του Ιουλίου, όταν όλοι θα υποβάλουν τις τροπολογίες τους και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, ώστε να βρούμε μια μέση οδό στην Επιτροπή μας. Η πρότασή μου η συνοπτική μπορεί να είναι η μέση πρόταση, όπως πάντοτε κάνουμε, αλλά για το κάνουμε αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε όπως κάνουν και οι ελείσες ε, στα ημερολόγια του πλοίου, γραπτός, με τις τροπολογίες μας. Ωραία. Έχουμε θέσει η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Η 28 Ιουλίου στις 12 η ώρα, άρα ο κύριος Γκάλαχερ και η κυρία Χιδέρο είπε, και ο κύριος Χάτον είπε να καθυστερήσουμε. Εσείς τι λέτε, θέλουμε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή ή να τα αφήσουμε στους συντονιστές για το απόγευμα. Mr. Gallagher, it's your proposal. Κύριε Γκάλαχερ, εσείς κάνετε την πρόταση. Γκάλαχερ. Δεν μου αρέσει που το λέω αυτό. Αν ήμουν στην Αδριατική, θα έλεγα εντάξει να προχωρήσουμε. Αλλά εμείς, εμείς είμαστε στην καρδιά του προβλήματος. Εγώ δεν θέλω να πιέσω κάποιον όταν πιέζεται. Δεν καταλαβαίνω. Αν είναι τόσο απλό, τότε αν δεν έχει επιπτώσεις, γιατί χρειάστηκε να γίνει συζήτηση. 2% είναι 2 ανά 100 άτομα. Είναι 2 άτομα. Είναι 2 άνθρωποι. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Φυσικά θα συζητήσω, θα συμφωνήσω με την ε, πλειοψηφία. Αλλά να, πούμε, να αποφασίσουμε σήμερα ή να το απορρίψουμε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο κ. Μιλάνα. Σίγουρα είναι κύριος. Ο κύριος Αρσένης. Ε, μα νομίζω ότι πρώτα ήθελε να μιλήσει η κυρία Ρόντουστ. Ευχαριστώ λέει η κυρία Ρόντουστ. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι κάνουμε πλέον σιγά σιγά. Εδώ έχουμε ε, απασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα αυτό. Είχαμε συμφωνήσει ως συντονιστέ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής τροπολογιών 8 Ιουλίου λοιπόν. Και τώρα πιστεύω ότι πρέπει να τηρήσουμε αυτή μας τη δέσμευση. Πρέπει κάποτε να καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί μας τελειώνει ο χρόνος. Έχουν συνεργαστεί τόσο πολύ, έχουν δουλέψει για το θέμα αυτό τόσο πολύ πρέπει εντός της παρούσας θητείας να λήξει το θέμα αυτό. Κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θέτει εν κινδύνο αυτό το στόχο. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, έχουμε εργαστεί τόσο πολύ, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία πλέον. Δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε τώρα, δεν το μάθουμε μέχρι 8 Ιουλίου. Πρόεδρος, να μην ξαναξεκινήσουμε τώρα συζήτηση. Παρακαλώ, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε παρακαλώ. Ποιοι θέλουν να τηρήσουμε την προθεσμία όπως έχει καθοριστεί. Οχτώ. Ποιοι θέλουν παράταση. Ένας. Σαφές. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών 8 Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει 18 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια θα γίνει στη δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 10. Η έκθεση του κυρίου Σαλαβράκου για την Μεσόγειο και τον Εύξηνο ο κύριος Σαλαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. I know everyone is exuberant after that uh, long debate, but a bit of silence. Ξέρω ότι είστε κουρασμένοι μετά από μια μακρά συζήτηση, αλλά παρακαλώ σιωπήστε λίγο μέχρι να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Λαμβάνω με την κόπο των συναδέλφων, διότι το θέμα που προηγήθηκε ήταν πολύ σημαντικότερο από αυτό το οποίο επακολουθεί. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος Πρώτον, ο ανταγωνισμός για τους ε, περιορισμένους αλλιευτικούς πόρους και τα θαλάσσια αποθέματα, όπως είναι γνωστόν σε όλους μας, έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η σχετική σπανιότητα των αλλιευτικών πόρων δεν είναι κάτι νέο, αλλά φαίνεται σήμερα να έχει ένα εγκευμένο φαινόμενο που επηρεάζει το θαλάσσιο υποσύστημα. Το πρόβλημα επιτείνεται από τους δημογραφικούς δείκτες. Σύμφωνα με έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Marine Policy το 2025 ο αστικός πληθυσμός στη Μεσόγειο θα έχει αυξηθεί κατά 60% διπλασιάζοντας τη ζήτηση για τα αλλιευτικά αποθέματα. Η Μεσόγειος είναι πιο στενή θάλασσα, δεν είναι Ατλαντικός όπως ξέρετε ε, και εκεί και ο ανταγωνισμός και τα αποθέματα είναι λιγότερα. Όπως φυσικά γνωρίζετε η διαχείριση της ελγίας και η θεσμοθέτησή της παρουσιάζει πολλές δυσκολίες σε σχέση με την ξηρά λόγω της κινητικότητας και της διακύμανσης των πόρων, της ποικιλία των τεχνικών αλληλείας και της ύπαρξης διαφορετικών καθεστώτων που διέπουν την πρόσβαση των σκαφών στην αλληλεία. Ενώ τα αποθέματα εξακολουθούν να μειώνονται, τα παράκτια κράτη φαίνεται να έχουν αποτύχει στην αποτελεσματική διαχείριση της αλληλείας. Στην έκθεσή μου γίνεται προσπάθεια απεικόνηση του προβλήματος και διατυπώνονται κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση συγκρούσεων που σχετίζονται με τις ελιευτικές ζώνες και τη διαχείριση της ελίας. Γίνεται ξεκάθαρο φυσικά ότι η βάση είναι η υπάρχουσα νομοθεσία, το διεθνές δίκαιο και κυρίως η σύμβαση του ΟΕ για τη θάλασσα, το δίκαιο της θαλάσσης, του UNCLOS. Είναι σαφές ότι τα χωρικά ύδατα και η διαχείριση των αλλιευτικών ζωνών αποτελεί υπόθεση που εμπίπτει στην εθνική δικαιοδοσία των κρατών. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι τα περισσότερα παράκτια κράτη της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας είναι τρίτα κράτη, είναι δύσκολο να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχοντας περιγράψει το γενικό πλαίσιο της έκθεσης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνο, μερικά, σε, μόνο σε μερικά σημεία που θεωρώ σημαντικά προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαχείριση τη αλληλείας και των χωρικών εδάτων στις λεκάνες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Πρώτον, πολιτική συνεργασία μεταξύ των κρατών. Η θαλάσσια διαχείριση στη Μεσόγειο και στη Μαύρη θάλασσα απαιτεί υψηλού επίπεδου πολιτική συνεργασία και συνοχή μεταξύ των παρακτήνων κρατών, καθώς και συντονισμένες προσπάθειες σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει δυσκολίες το πρώτο. Το άρθρο 23 της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών που βρίσκονται σε κλειστές, σε enclosed μερικώς σε μη enclosed θαλάσσιες δακάνες. Όπως είπα υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει διαφορετική κουλτούρα κρατών, υπάρχουν τρίτα κράτη τα οποία ε, ακόμη δεν έχουν ε, φτάσει σε κάποιο επίπεδο ε, εκμοντερνισμού του τρόπου της αλληλείας κτλ πρέπει να υπάρξουν διμερείς συμφωνίες. Δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη της θαλάσσης αυτής δεκανής είναι τρίτα όπως είπα, δεν υπάγονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, είναι μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα το να φτάσουμε σε διμερείς συμφωνίες και πρέπει να ενισχυθούν ώστε έτσι να μπορεί να εξασφαλιστεί μια χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση στις περιοχές αυτές. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασφάλιση του σεβασμού των κανόνων η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του διπλωματικού της, ε, της διπλωματικής της για τη διασφάλιση του σεβασμού των κανόνων, των αρχών και της ευρωπαϊκής κοινωνικής ελληνικής πολιτικής και του διεθνούς δικαίου, ειδικότερα σε σχέση με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες που πρέπει να συμμορφωθούν και να σεβαστούν το κοινοτικό κεκτημένο. Σημαντικός κρίνεται ο ρόλος του GFMI C της Γενικής Επιτροπής Ελίας για τη Μεσόγειο για τη διασφάλιση βιώσιμης ελίας και των ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Η σύμβαση UNCLOS. Από τα 21 μεσογειακά κράτη μόνο τρία δεν έχουν υπογράψει ή επικυρώσει τη σύμβαση του ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Το Ισραήλ, η Συρία και η Τουρκία. Δεδομένου όπως προελέχθη ότι η σύμβαση αυτή είναι μέρος του διεθνούς δικαίου και της ευρωπαϊκής νομολογίας, για τη διαχείριση των υδάτων και των αλλιευτικών πόρων θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει διπλωματική πίεση μέσω των εργαλείων της κυρίας Άστον ούτω ώστε να προχωρήσουν και οι χώρες αυτές στην υπογραφή της συμβάσεως αντλος, ε, ειδικότερα ε, σε χώρες που βρίσκονται υπό ενταξιακό καθεστώς σήμερα διότι το να ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε αυτή την εποχή της Συρία να έχουμε κάποια αποτελέσματα δεν το βλέπω και θα ήμουν εκτός πραγματικότητας. Τέλος, ε, η θαλάσσια διαχείριση, η προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος και των αλληλευτικών πόρων καθώς και ο έλεγχος για την παράνομη άναρχη και λαθρέα ελιέ την ΑΙΓΙΟΥΙΟΥ έχει αποδειχθεί ότι προστατεύεται καλύτερα όταν υπάρχει ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο Κατά αυτόν τον τρόπο, μέσα από την εκθεσή μου ενθαρρύνει τη δημιουργία θαλασσίων ζωνών και ειδικότερα η ανακήρυξη αποκλειστικών οικονομικών ζωνών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως και καλείται η Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο να συνδράμει στον τομέα αυτό παρέχοντας καθοδήγηση και την ανάλογη υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Σημειώνω μόνο έξι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε λίγο θα είναι 7 λόγω ένταξη της από τα 22 κράτη Μεσογείου είναι παράκτια αν αυτά τα έξι ή εφτά μετά από λίγο κράτη-μέλη ανακήρυξαν ΑΟΣ, θα, ήλεγχαν, θα ελεγχόταν από πλευράς ευρωπαικη Ένωσης περίπου το 60% των χωρικών υδάτων της Μεσογείου με αποτέλεσμα ε, και οικονομικό και κοινωνικό για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της εκθέσεως. Δεν θέλω να σας κουράσω παραπέρα. Θα ακούσω τις ε, απόψεις των συναδέλφων, τις οποίες θεωρώ και χρήσιμες και επικοδομητικές και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερος κύριε Σαλαβράκο. Η κυρία Μάσνα. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Σαλαβράκο για την έκθεσή του. Όντως, στην Μεσόγειο και τον Εύξηνο η υπεραλίευση είναι μεγάλο πρόβλημα, έχουν μειωθεί κατά πολύ τα αποθέματα και υπάρχει πίεση, οι αλληλείς ε, δεν μπορούν να ε, αλλιεύσουν επικερδώς. Είναι πρόβλημα αυτό και προκαλεί συγκρούσεις. Όπως υπόθηκε, δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη της περιοχής ε, μέλη της Ένωσης, αυτό δεν διευκολύνει τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει διάλογος και εκτός των ορίων για να λύσουν τα προβλήματα. Ο διμερής διάλογος είναι μια καλή βαριάντα και παράλληλα η σύμβαση ένκλος ε, είναι γνωστό, δεν έχει επικυρωθεί από όλους. Βεβαίως θα ήταν επιθυμητό, αλλά το θέμα είναι υπάρχει καμία δυνατότητα να τους ε, υποχρεώσουμε. Θα πρέπει να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των ε, αποθεμάτων, όπως και παντού αλλού, αλλά μόνο εάν συνεργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Οι προτάσεις του ζυγητή νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και εάν καταφέρουμε να υπάρξει βιώσιμη αλληλεία στις περιοχές αυτές, αν συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση, τότε θα συμβάλλουμε στην εκπλήρωση των στόχων της ε, κοινή ελευτικής πολιτικής και πέραν των συνόρων μας, αυτό θα ήταν σκόπιμο. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω σε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Λαβράκο για την έκθεσή του. Νομίζω ότι οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. η αλληλεία μας ενδιαφέρει σε όλες τις περιοχές, Βαλτική, Ατλαντικός, ε, Μεσόγειος. Έχουμε επιτύχει μια ενοποιημένη προσέγγιση. Χαίρομαι που η Κομισιόν έκανε μια εκτίμηση τι αποθέματα υπάρχουν στα βόρεια τμήματα των ε, θαλασσών, ούτως ώστε να υπάρχει ε, βιώσιμη αλλήλευση. και είπαμε ότι δεν πρέπει να υπερβληθεί το 60%. Βεβαίως θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και πρέπει και στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο να ισχύουν οι ίδιες αρχές. Και εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτύχουμε μέσω διαπραγματεύσεων, διότι οι μη χώρες μέλη είναι η πλειονότητα. Εμείς βέβαια έχουμε τη βόρεια πλευρά της Μεσογείου και έχουμε διαπιστώσει για παράδειγμα ότι στη σύμβαση για τον τόνο οι Αιγύπτιοι και οι Σύροι επίσης ενδιαφέρονται, αλλά και άλλες χώρες της Βόρειας Αφρικής έχουν άλλους στόχους και είναι πολύ περίπλοκη η επίτευξη στόχων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο η διπλωματική οδός. διμερεί συμφωνίες επίσης πρέπει να συναυθούν, η μία μετά την άλλη. Αυτό ισχύει και για τον Εύξηνο. Ε, Τουρκία, Ουκρανία, Ρωσία πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Πρέπει και οι δικοί μας αλλοίς να τηρούν τις, ε, ε, τους κανόνες, αλλά αυτό δεν πρέπει να τους οδηγεί σε μειονεκτική θέση. Και παράλληλα πρέπει να ε, προστατεύουμε τα αποθέματα. Γι' αυτό κεντρικό είναι και σε αυτές τις διμερείς διαπραγματεύσεις να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε να υπάρχουν και να διεξάγονται έλεγχοι. Όχι μόνο επί των δικών μας αλληλείων, οι έλεγχοι αυτοί να μπορούν να ελέγχουν τα σκάφη, να βλέπουν τι έχουν αλλιεύσει, ε, αν παραβιάζουν τις συμφωνίες κτλ. Χωρίς έλεγχο δεν πρόκειται να ισχύσει τίποτα, να εφαρμοστεί τίποτα και βέβαια είναι δυσχερής ο έλεγχος. Πρέπει όμως οπωσδήποτε να το δούμε το θέμα αυτό, γιατί σχετίζεται και με την εξωτερική μας πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σαλαβράκο που έκανε μια καλή ανάλυση της κατάστασης. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Ο κύριος Μιλάνα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Σαλαβράκο που συνόψισε νομίζω αρκετά καλά ε, όλα τα θέματα. Κάποια σημεία μόνο θέλω να υπογραμμίσω. Καταρχήν αυτό τη διμερούς συνεργασία με τα άλλα κράτη που είναι σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω πω ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε μια πραγματική πολιτική συμφωνιών ε, αλληλευτικών με αυτές τις χώρες. Και το λέω πολύ απλά και ξεκάθαρα. Μια λεκάνη όπου βρέχονται 8 κοινοτικέ χώρε και 22 μη κοινοτικέ, έχει τα 2 τρίτη των ακτών χωρί έλεγχο από πλευρά των ευρωπαϊκών αρχών. Δεν υπάρχει πολιτική που να μπορεί να την εφαρμόσει. Εάν δεν φτιαχτεί πραγματικά με στρατηγικό τρόπο μία σχέση αλλιευτικών συμφωνιών που θα ξεπερνούν τις διμερείς σχέσεις πολιτικού επίπεδου με τις χώρες αυτές. Χρειάζονται αλλιευτικές συμφωνίες και αυτές μπορεί να είναι δαπανηρές για την Ευρώπη. Μπορεί να είναι δαπανηρές δηλαδή. Είναι χρήματα όμως τα οποία θα δαπανηθούν καλά, ε, ιδιαίτερα προς κάποιες ε, αφρικανικές χώρες, για να έχουμε και περισσότερο έλεγχο. Αυτό είναι πρώτη, το πρώτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω. Το δεύτερο είναι η μη εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο. Δεν εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός. Οι επιπτώσεις αυτού του κανονισμού είναι... Και κοιτάξτε, δεν εφαρμόζεται σε ένα βαθμό λόγω προσεξίας των κρατών μελών, ε, σε ένα βαθμό λόγω αδιαφορίας του τομέα και τρίτον γιατί δεν ήταν καλός. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος να το πούμε γιατί δεν ε, είναι σωστά. Εξάλλου, ο κανονισμός προέβλεπε τον Ιούνιο του 2013, δηλαδή τώρα, να ξεκινούσε το τμήμα από πλευράς μάλλον της Κομισιόν η επαλήθευση του εφαρμογή. Ας το κάνει. Ας το κάνει και γρήγορα. Και μάλιστα θα ήθελα να ε, αναφερθώ στην, αρχή, στην νομική αρχή που προβλέπει την επαλήθευση της εφαρμογής του κανονισμού για τη Μεσόγειο τον Ιούνιο του 2013 και έπειτα. Η διαχείριση της θάλασσας η ίδια. Εμείς έχουμε μια προσέγγιση που είναι βασικά σε αυτή την θάλασσα, που είναι κλειστή θάλασσα βασικά, όπου, και αυτή τη φράση την έχω πει, είναι ένας χώρος όπου μπορούμε να κάνουμε αναλήψεις και η δραστηριότητα την οποία κάνουμε είναι να περιορίζουμε τις αναλήψεις μέσω κανόνων κανόνων λιγότερο ή περισσότερο περιοριστικών. Μα δεν είναι μια θάλασσα ε, για την οποία μπορεί να εφαρμόζεται αυτή η αρχή. Είναι μια θάλασσα που πρέπει να μετατραπεί πολιτικά σε ένα μεγάλο ε, ε, κάμπο που θα πρέπει να τον καλλιεργήσουμε γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε καμία θετική διέξοδο και θα πεθάνει, θα νεκρωθεί η θάλασσα αυτή. Πρέπει να επανέλθουμε στην αρχή του και να καταλάβουμε πώς πώς θα γίνει μια μεταρρύθμιση ώστε να μπορέσουμε πολύ στοχευμένα να εσωματωθεί ε, η υπόθεση των ε, κλειστών περιοχών. Εγώ δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά η ιδέα του να καλλιεργηθεί η ε, Μεσόγειος και ο εύξηνος πόντος αντίθετα από το τι μπορεί να γίνει στον Ατλαντικό είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι μπορούμε να προσανατολίσουμε διαφορετικά τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και τελευταίο θέμα, δεν υπάρχει χώρο στην Ευρώπη πιο κατάλληλος για να υλοποιηθούν ε, μορφές ε, ε, θαλάσσιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Αν ξεκινήσουμε από τον χώρο αυτό, είναι ζωτική σημασία για τη Μεσόγειο και το γεγονός ότι πρέπει να σχεδιαστούν οι περιοχές, οι ζώνες, δηλαδή να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και από τις έξω, χώρες να δείξουν τους χώρους, να υποδείξουν πού γίνεται η αλληλεία, πού γίνεται ο τουρισμός, πού γίνονται μεταφορές, στη θάλασσα της Μεσογείου, γιατί αυτό είναι η σωτηρία της Αλίας. Σκεφτείτε ότι μόνο στα ύδατα, μάλλον εντός των 40 μιλίων, δηλαδή πέρα από τα χωρικά ύδατα, στη χώρα μου υπάρχουν 1.200 πλατφόρμες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, οποιασδήποτε απόφασης μιας πετρολοβιομηχανίας που αποφάσισε να επενδύσει στην τάδε μεριά. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το αφήνουμε να συνεχίζεται. Μπορεί να είναι αντικείμενο όπου η Κομισιόν απλά και μόνο παρακολουθεί ως απλός θεατής ή θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου ο σχεδιασμός θα είναι το μέσο δια του οποίου θα υπάρξει συγκεκριμένος προγραμματισμός. Εγώ θα κάνω κάποιες ε, ε, τροπολογίες που θα είναι σχετικές με τις θέσεις για κάποιες διορθωτικές μικρές, κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις. Λοιπόν, για αυτά που σας είπα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αρσένης. Πρόεδρε, Καταρχήν ε, να ενώσω τη φωνή με τους συναδέλφους που συνεχάρισαν τον εισηγητή ε, για την εξαιρετική του δουλειά και την ε, μετριοπαθή και μετρημένη στάση στο, στο ζήτημα πιάνοντας όλα τα κρίσιμα σημεία. Τα θέμα, το θέμα που συζητάμε είναι ένα θέμα που οι ψαράδες στη Μεσόγειο αντιμετωπίζουν καθημερινά. Είναι η η μη εφαρμογή της, ε, η μη κοινή υπογραφή και αποδοχή των αρχών της Ούγκλος, ε, αλλά και η έλλειψη συμφωνίων διαχείρισης μεταξύ γειτονικών χωρών ε, που πολλές φορές οδηγεί σε δυσκολίες στους ψαράδες που μπορεί να φτάσουν μέχρι και απειλή της ζωής τους και πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει λόγος να μην βρεθεί μια λύση σε αυτό. Μπορούμε να βρούμε μια λύση. Νομίζω ότι και οι ιδέες του κυρίου Μιλάνα αναφορικά με, τις, ε, με τη δυνατότητα να γίνουν αλληλευτικές συμφωνίες ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αναφέρουμε στις ιδέες κιόλας του κ. Μιλάνα και της Ρίας Ρόντους που υποστήριξαμε όλοι μας στα πλαίσια της ΕΦΤ για συμφωνίες αλληλευτικές χωρίς αντικείμενο την, αλη, την ε, με αντικείμενο την ε, υιοθέτηση από γείτονες χώρες των κοινών κανόνων είναι πράγματα που πρέπει να, το, τα, εξετάσουμε. Ε, θα στηρίξω όλες τις καλές ιδέες που ε, ακούστηκαν και την εισήγηση του συγκητή και πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει ακόμα περαιτέρω προσοχή στο ζήτημα. Ε, είναι ένα ζήτημα από το οποίο εξαρτάται και η ευημερία και πολλές φορές και η ειρήνη. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με, την αίσθηση του επίγοντος. Ευχαριστώ. Κυρία Λέβεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Σολαβράκο, γιατί πραγματικά η έκθεση είναι εξαιρετική και καλύπτει σχεδόν όλα τα θέματα. Μεγάλη πρόκληση η διαχείριση μια θάλασσα από την οποία βρέχονται και κοινοτικέ και εξωκοινοτικέ χώρες. Για δεκαετίε ολόκληρε είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα και στη Βαλτική. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διαχείριση των ελευτικών πόρων, ενώ μερικέ χώρες ανήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες όχι. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να υπολογίζουμε ε, στην ε, προσχώρηση όλων των ε, χωρών της Μεσογείου ή της Μαύρης Θάλασσας στην προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε στη Βαλτική. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε τις συμφωνίες για τη σωστή διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Έχουμε τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι σημαντικό υπογράφοντες να ενστερνίζονται αυτέ τι αρχέ για να γίνεται σωστή η διαχείριση των ολιστικών πόρων, μεταξύ άλλων και τη αρχή τη μέγιστης βιώσιμη απόδοση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το θέμα τη ΦΑΟ. Έχω μάλιστα και την Ειδική Επιτροπή της Μεσογείου. Οπότε όλες οι χώρες θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στις διεθνείς τους υποχρεώσεις, γιατί στο κάτω-κάτω έχουν υπογράψει διεθνείς συνθήκες που διέπουν τη διαχείριση και θα πρέπει ε, να προβαίνουν σε αυτή τη χρηστή διαχείριση των αλληλευτικών πόρων. Στο σημείο 7 ε, αναφέρει ο κ. Σαλαβράκος τη χρήση των διπλωματικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει πίεση σε τρίτε χώρε να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και στη συνέχεια, στην παράγραφο 8, επισημαίνεται το γεγονός ότι υποψήφιες για ένταξη χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν τη συμφωνία Άγκλος και να γίνουν μέλη δηλαδή αυτής της συμφωνίας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα και κάποια υποψήφια χώρα θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά, ότι πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να κυρώσει τη συμφωνία ή συνθήκη για το δίκαιο της θάλασσας. Στο σημείο 8 αναφέρεται ότι Μόνο τρεις χώρες δεν έχουν υπογράψει την Άγγλος, τη συμφωνία του ΟΗΕ. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές οι τρεις χώρες. Νομίζω ότι προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ε, και την Περιφερειακή Επιτροπή Ελίες, κάτι που απαιτείται ήδη. Σας ευχαριστούμε κυρία Λόβιν. Έχουμε την κυρία Παρία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του που πραγματικά είναι εξαιρετικής ποιότητας και συνοψίζει με πολύ εύστοχο τρόπο τα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη Μεσόγειο και στον Εύξηνο Πόντο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως ε, τις παρατηρήσεις σας και όλοι συμφωνούμε ως προς το δυναμικό ανάπτυξης ε, της Μεσογείου. Αυτό θα πρέπει να διαφυλαχθεί και οι συγκεκριμένες προκλήσεις ε, θα έχουν ευρελεγγύη σημασία για το σύνολο της περιοχής. Σε ό,τι αφορά την ε, βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Μεσογείου προκειμένου να αξιοποιηθεί το οικονομικό δυναμικό με βάση τους ελευτικούς πόρους, Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό και διοικητικό πλαίσιο που θα είναι κατάλληλα, μια χρηστή διακυβέρνηση και ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης πόρων που θα συνοδεύεται από ένα σύστημα ελέγχου και σεβασμού των ελεκτικών μέτρων που θα έχει συμφωνηθεί ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριο Μιλάνε για την εφαρμογή του κανονισμού για τη Μεσόγειο, εγώ δεν θα ήμουν τόσο κατηγορηματική. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Βέβαια, συμφωνώ ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας, αλλά εδώ και μία-δύο τριετία έχουμε λησαλέο αγώνα ε, απέναντι στα κράτη-μέλη που κολυσιεργούν και δεν εφαρμόζουν ακόμη τον ε, κανονισμό. Έχουν υιοθετηθεί πάντως διάφορα σχέδια δράσης από κράτη-μέλη και έχουν εφαρμοστεί. Σε αντίθετη περίπτωση ξεκινούμε διαδικασία επιπαραβάση κατά των χωρών που δεν ε, εφαρμόζουν τον κανονισμό και σίγουρα έχουμε και πιο αυστηρούς ελέγχους ως προς το θέμα αυτό. Και ναι, μεν, ε, Αργήσαμε κάπως, αλλά σίγουρα την τελευταία τριετία έχουμε σημειώσει πρόοδο. Όπως επισημάνατε πολύ εύστοχα, οι περισσότερε από τι χώρε που βρέχονται από τη Μεσόγειο δεν είναι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η ανάγκη στενή συνεργασία με τι χώρε αυτέ. Και σε διμερές επίπεδο, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω την ανάγκη μιας συνεργασίας στα πλαίσια των ε, υπαρχών των οργανισμών ε, και φόρουμ της Μεσογείου, είτε στην Γενική Επιτροπή Αλίας της Μεσογείου, και θα αναφερθώ πιο λεπτομεριακά σε αυτό, αλλά και στα πλαίσια του ICAT. Γιατί ο ICAT έχει θεσπίσει δρακόντια μέτρα σε ό,τι αφορά κάποια πελαγικά είδη της Μεσογείου, ιδιαίτερα τον ερθροτόνο αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη δρέψει τους καρπούς αυτής της αυστηρής πολιτικής ε, στην οποία πρωτοστατήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε και οι πρώτοι που την εφαρμόσαμε. Και οι συνθήκες Βαρκελόνης ε, και Βουκουρεστίου για, την, για τον εύξηνο πόντο είναι σημαντικές και την σύμβαση ΑΚΟΜΠΑΜΣ για τα ΚΙΤΗ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και στα πλαίσια της ε, CGPM εδώ και δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια έχουμε μια πολύ ενεργό πολιτική προκειμένου να εφαρμόσουμε ε, διαχειριστικά σχέδια ώστε να συντονιστούν ε, οι διάφοροι φορείς της κοινή ελευθερικής πολιτικής στη Μεσόγειο. Και μάλιστα για πρώτη φορά έχουμε και για τα μικρά πελαγικά είδη της Αδριατικής για πρώτη φορά ε, σχέδιο διαχείρισης και επίσης για πρώτη φορά έχουμε τεχνικά μέτρα για τον εύξηνο πόντο. Ας μην τα ξεχνούμε όλα αυτά και ας μην ξεχνούμε επίσης ότι προωθούμε μία ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση του CGPM προκειμένου να εξασφαλίσουμε συνθήκες θεμητού και ίσου ανταγωνισμού και μια γενική πολιτική εδώ. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, έχουμε ξεκινήσει διάλογο για αλληλευτικά θέματα με την Τουρκία, την Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο διάλογος αυτός ε, είναι μεν χρονοβόρος, αλλά τουλάχιστον ε, είναι υπαρκτός. Και θα το συνεχίσουμε, ε, όπως θα συνεχίσουμε και το διάλογο με τις χώρες της Νοτίας Όχθης της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά το δίκαιο για την, τη συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, η προσέγγιση για τα σημεία αυτά είναι ευκταία και εύλογη και όπως είπατε η διεύρυνση των οικονομικών αποκλειστικών ζωνών αποτελεί αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα και όχι κοινοτική. Πάντως πριν από λίγα χρόνια εκπονήσαμε μελέτη για τα πλεονεκτήματα των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Έχει ολοκληρωθεί πια η μελέτη αυτή και θα γίνει επίσημα και η παρουσίασή της ε, στο εγγύς μέλλον από την Αρμόδια Επίτροπο. Γίνεται μια, γίνονται διάφορες προτάσεις για πρωτοβουλίες προκειμένου να προωθηθούν αυτές οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και στη Μεσόγειο για τις χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμη δηλαδή. Για όλες τις χώρες ε, της Μεσογειακής Λεκάνης. Επίσης, να πω δύο λόγια για την επιστημονική συνεργασία, κάτι που επίσης αναφέρατε στην έκθεση. Η επιστημονική συνεργασία είναι νευραλική σημασία και απολύτω απαραίτητη για να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένη άποψη για την κατάσταση των αλευτικών ε, αποθεμάτων και να χαράξουμε την πολιτική διαχείριση. Και εδώ και χρόνια έχουμε κοινά σχέδια με τη ΦΑΟ με συμμετοχή μεσογειακών χωρών, τα, τα σχέδια ISMED, COPEMED, SUDMED, όλα αυτά τα σχέδια και προγράμματα στόχο έχουν τη βελτίωση της επιστημονικής συνεργασίας σε όλες τις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της έκθεσής σας. Τη χαιρετίζουμε με ενθουσιασμό και θα συνεχίσουμε να προωθούμε το διάλογο με τις τρίτες χώρες προκειμένου να ενισχυθεί η διαχείριση των αλληλευτικών πόρων στη Μεσογειακή Λεκάνη. Και είμαστε φυσικά και υπέρ της συνεργασίας μαζί σας για την επιτεύξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Παριά. Και τον τελικό λόγο φυσικά θα τον έχει ο εισηγητή μα, ο κύριος Αλαβράκο. Ε, ευχαριστώ όλου του συναδέλφους και την Επιτροπή για την θέση που έλαβαν απέναντι στην εκθεσή μου. Επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόποση στα μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο ίσως αναζωπηρώσει τη διάθεσή σας. Ξέρετε πού οφείλει αυτό το κράτος, το Βέλγιο, στο οποίο ζούμε, ε, το γεγονός ότι απεκόμισε πολύ πλούτο σε ένα νομικό παράδοξο. Ανεγνώρισε την εταιρεία εκμετάλλευσης Κονγκό ως κράτος. Ανεγνωρίστη με τις σύμβαση του Βερολίνου είναι το μοναδικό φαινόμενο που υπάρχει στη διεθνή ιστορία που ανεγνωρίστη σαν κράτος μια ανώνυμη εταιρεία. Η εκμετάλλευση του Κονγκό έδωσε τον πλούτο στην ε, ή ε, στο κράτος αυτό το οποίο ζούμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι όλες οι αυτοκρατορίες που έγιναν στην Ευρώπη ιστορικά και διεθνώς βασίζονται όχι μόνο στην ισχύ αλλά και στο εμπόριο, στην κατοχήρωση εμπορικών σχέσεων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάμαι ότι έχει ένα πρόβλημα. Η εταιρεία των ε, ε, η Επιτροπή Οικονομικών, ο Επίτροπος Οικονομικών, ο Επίτροπος ε, Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Επίτροπος Ελίας, ο κάθε Επίτροπος δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Γιατί. Δίνουμε στην Αίγυπτο 5 δισεκατομμύρια ευρώ βοήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε κάνε διμερείς συμφωνίες διότι σου δίνουμε αυτή τη βοήθεια η οποία είναι σημαντική και είναι και δωρεάν με τα παράκτια λοιπά κράτη εις τρόπον να υπάρχει μια εκμετάλλευση, μια ομαλή εκμετάλλευση των αλλιευτικών πόρων, των, ε, πόρων ε, σε διάφορους είδους δραστηριότητες κτλ. Και αυτό είναι μέσα στο θεμητό ανταγωνισμό και εμπόριο μεταξύ των κρατών που το χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί το 2025 όπως ξέρετε θα είμαστε περίπου από 8 που είμαστε του παγκόσμιου πληθυσμού θα είμαστε γύρω στο 5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Και χρειάζεται να έχουμε πόρους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πόρους για τα παιδιά μας. Το λέω αυτό ε, απλώς για να προβληματίσω πέραν της εκθέσεως και για άλλες ε, σχέσεις, συνοδευτικές σχέσεις και δράσεις τις οποίες μπορεί να κάνουν οι επίτροποι μεταξύ τους και εμείς με τους επιτρόπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Λυπάμαι που δεν υπήρξε χρόνος για την έκθεση της κυρίας Γκουτιέρδεθ για τις γυναίκες. Λυπάμαι ότι θα πρέπει να περάσει ως τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη γιατί δεν μπορούμε να υπερβούμε το χρόνο μας. Η συνεδρίαση των συντονιστών θα γίνει στις 3. Θα τα πούμε λοιπόν στις 3. Και η προθεσμία η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι στις 12 το μεσημέρι στις 24 Ιουνίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου και θα περάσει στην Ολομέλεια, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Τρεις η ώρα παρακαλώ για τους συντονιστές. Ευχαριστώ.